Right, um, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Συγκεντρώθηκε η απαρτία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκρισή της. Μπορούμε να την εγκρίνουμε παρακαλώ. Έχω μερικές ανακοινώσεις. Καταρχήν το άτυπο εκοφήν στη Λευκοσία. Το παρακολούθησα ως πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ, γιατί τώρα τακτικά μας προσκαλεί το ΕΚΟΦΗΝ. Στο κυρίω θέμα ήταν η Τραπεζική Ένωση και η κρίση του δημοσίου χρέους. Και εγώ παρουσίασα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τραπεζική Ένωση και τις κοιόδης τραπεζικές υπηρεσίες, μια και έχουμε πια διαμορφωμένη θέση για τα ζητήματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά του τριμερείς διαλόγους για το CRA3, Στι 13 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα ο τρίτος τριμερείς διάλογος, ε, υπερβολική έκθεση, δημόσιο χρέος και στοιχεία του συζητήθηκαν. Μέχρι το τέλη της εβδομάδας θα εξεταστούν οι συμβαστικές τροπολογίες και θα συνταχθεί ένα ανεπίσημο έγγραφο για την αστική ευθύνη. 27 ε, Σεπτεμβρίου είναι ο επόμενος τριμερής διάλογος. Το 7ο τώρα στατιστικό πρόγραμμα. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε υπό την προεδρία του Έντουαρτ Σικλούνα, που είναι και εισηγητής για το θέμα αυτό και καλύφθηκε το νομοθετικό σκέλος ε, βρέθηκε συμφωνία για πολλά θέματα, βέβαια κρεμούν κάποια. Το παράρτημα θα συζητηθεί σε επόμενο τριμερή διάλογο που κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα στις αρχές Οκτωβρίου για το CRD4-CRR, τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Θα συνεχιστούν τα έχιστα εργασίε το Σεπτέμβριο. Έχουμε δύο συμβαστικέ προτάσει για μηχανισμού κεφαλαίου και ε, τι μειώσεις και του ομίλου τραπεζών. Βέβαια, η συνολική πρόοδος ήταν μάλλον αργή και στις 11 Σεπτεμβρίου, στον τελευταίο πολιτικό τριμερή διάλογο, τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με την κατάσταση αυτή και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς δεσμεύσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Βασιλείας 3 στις αρχές του 2013. Βέβαια έγιναν κάποια σχόλια και από τα άλλα θεσμικά όργανα ε, κατηγορώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αργή πρόοδο και μάλιστα για να δηλώσει τον τύπο, πολύ άδικες και ανακριβείς, γιατί δεν είχαμε εντολή από τα άλλα δύο μέρη του εταίρους μας στην τριμερή διάλογο. Και χωρίς διαπραγματευτική εντολή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Αυτά για το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τώρα το διπλό πακέτο, τρίτος τριμερής διάλογος. Χθες 18 Σεπτεμβρίου είχαμε τους δύο, τη συζήτηση των δύο κανονισμών ανά άρθρο. Έγινε κάποια πρόοδος, αλλά έμειναν αρκετά θέματα έκρεμοι. Οπότε θα συζητηθούν στον επόμενο τριμερή διάλογο που θα λάβει χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου, 3 με 6.30. Για το Omnibus. Χθες είχαμε τον ένατο τριμερή διάλογο για το δεύτερη συμφωνία Omnibus. Προτάθηκε από τον, κύριο, από τον Επίτροπο Μπαρνιέ ε, τεχνική αξιολόγηση που θα πρέπει να γίνεται εξάντε για τις μακροπρόθεσμες εγγύησεις προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα γίνει και τεχνική αξιολόγηση με έκθεση που θα δημοσιευθεί το Μάρτιο του 2013, κάτι που προϋποθέτει τη συνέχιση τότε των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει γραπτή δήλωση για τις συνέπειες αυτής της πρότασης κατά την προκαταρκτική εκτίμηση και την καθυστέρηση που θα προκαλέσει. Πρώτα θα εξεταστούν οι προτάσεις και μετά θα μας ενημερώσει για την πορεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, στα σημεία 15 και 16 της ημερήσιας διάταξης θα αντιστραφούν μετά από αίτηση της εισηγήτριας ε, για τις ποινικέ κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Πρώτα θα συζητηθεί το 16. Αυτά. Δηλαδή, τις ποινικέ κυρώσεις και την κατάχρηση αρμοδιοτήτων στην αγορά θα τις συζητήσουμε πριν την έκθεση για την ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Μία αντιστροφή λοιπόν το σημείο 15 και 16 όπως σας είπα. Αυτές είναι οι αλλαγές. Ο κύριος Λάγκεν. Κυρία Πρόεδρε, έχω μία ερώτηση. Πότε έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του Ιβμέρς. Α. Συγγνώμη, Βέρνερ, δεν φοράω τα ακουστικά μου. Ε, αγγλικά πρέπει να μιλάμε συνέχεια. Κάντε και κάνα μάθημα. Κάνα γαλλικό, γερμανικό. Με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, έχω μία ερώτηση. Πότε έχει προγραμματιστεί η ακρόση του Ιβμέρς. Έχω λάβει μία πρόταση. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πριν τη, την άτυπη. Γιατί μην ξεχνάτε πως η πρόταση υπάρχει εδώ και τρεις ή μισή μήνες. Um, για ποια πρόταση είπες? Την ε, πρόταση του κυρίου Κοζές. Ακρόαση του Ιβ Μέρς. Πότε θα γίνει, πότε προβλέπετε ή τι πρόγραμμα έχουμε. Ε, Θα σε ενημερώσω. Όπως ξέρεις, συναντήθηκα με τον Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη για την ακρίβεια, και μάλιστα ενημέρωσα σχετικά τους συντονιστές. Ε, στη συνέχεια ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα συζητήθηκε και στη διάσκεψη των πρόεδρων και κατά τη γνώμη μου ε, θα υπάρξει κάποια επικοινωνία του πρόεδρου Σούλτς με τον πρόεδρο του Eurogroup αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια ανακοίνωση. Δεν με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μου είπε ότι περίμενε μια τέτοια επικοινωνία με τον πρόεδρο. Αυτό μου το είπε στην Λευκοσία. Γνώρι, ε, ρώτησα τη γραμματεία, αλλά από ό,τι ξέρω πρόοδος δεν υπάρχει για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν έχει διευθετηθεί. Δεν άλλαξε η θέση της Επιτροπής μας πάντως, μετά την τελευταία συζήτηση των συντονιστών της περασμένης Τρίτης το πρωί. Και μάλιστα τότε οι συντονιστές που εκπροσωπούσαν την πλειοψηφία εξέφρασαν την ικανοποίησή τους. Δύσκολο βέβαια αυτό, μια και δεν έχουμε πληροφορίες και δεν ξέρω αν μπορούμε να διοργανώσουμε την ακρόαση, γιατί υπάρχει και ανάμειξη της διάσκεψης των Προέδρων. Πάντως, αν συμφωνήσουμε, μπορούμε να την οργανώσουμε, ώστε να ψηφίσουμε τον Οκτώβριο. Προσωρινά πάντως, η Γραμματεία είπε ότι μπορούμε στις 26 Οκτωβρίου να την οργανώσουμε, αν μέχρι τότε έχουν διευθυνθεί τα πράγματα. Αυτά ξέρω εγώ. Επίσημα πάντως, δεν έλαβα καμία απάντηση από κανέναν. Μετά τη συνάντηση που είχαμε τον Ζαγκλοντ Τζουνκέρ την περασμένη Τρίτη. Κύριος Γκοζές, ευχαριστώ και ευχαριστώ που απαντήσατε στο mail που σας έστειλα. Ε, επιβεβαιώνω εδώ την θετική στάση του ΕΛΚ και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και γυναίκες στη διαδικασία επιλογής ε, των στελεχών των διαφόρων οργανισμών. Ό,τι έγινε έγινε, ό,τι έπρεπε να γίνει μάλλον έγινε και τώρα καλούμαστε να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να ε, διακόψει ή να καθυστερήσει την ακρόαση με τον κύριο Μέρς που εντάσσεται στην κανονική διαδικασία που προβλέπουν οι συνθήκες. Το άρθρο 283 της συνθήκης προβλέπει ε, μία πρόταση του Συμβουλίου, μία υποψηφιότητα για την οποία καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό και το είπα στους συντονιστέ είναι ότι η διαδικασία που προηγείται της, του διορισμού λαμβάνει υπόψη και την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβω μια απόφαση και όχι να εφαρμόσουμε κανόνες αντιφατικούς με τη συνθήκη. Πάντως, επειδή θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, θεωρώ ότι είναι εκνευριστικό, ενοχλητικό να θεωρήσει κανείς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εργή στο διορισμό ενός μέλους της ΕΚΤ, ενώ βρίσκεται η ΕΚΤ στο επίκεντρο με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει και τη θέση που θα έχει στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης. Γι' αυτό και ζητώ να διοργανωθεί το συντομότερο δυνατό η ακρόαση με τον κύριο Μπέρς. Και δεδομένου ότι μπορούμε να ψηφίσουμε στις 26 Οκτωβρίου, νομίζω ότι αυτή θα ήταν η σωστή διαδικασία. Πάντως, ε, καταλάβατε πολύ σωστά τη θέση μου και σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν ε, με ρώτησαν ε, τα μέσα ενημέρωση, ε, ξεκαθάρισε ότι καταλαβαίνω και τη δική σα θέση και του ΕΛΚ. Αλλά ακόμη δεν είχαμε ανταλλαγή απόψεων με άλλου συντονιστέ. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλη συζήτηση για το θέμα αυτό. Αλλά αν θέλετε να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο, ευχαρίστω. Αστρίτ. Ναι, Πρόεδρε. Είπατε ότι η ακρόση θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν είχαν επιληθεί κάποια ζητήματα. Τουλάχιστον αυτό άκουσα εγώ από τη μετάφραση. Μπορείτε να μου πείτε, δηλαδή, τι πρέπει να ρυθμιστεί ακριβώς. Όπως σας είπα, περιμένουμε κάποια ανταλλαγή ενημέρωσης. Νομίζω ότι το θέμα της ισότητας των φύλων να τα ξαναπώ από την αρχή. Το θέμα της ε, ισορροπίας ε, ε, των δύο φύλων, συζητήθηκε στη Λευκοσία και νομίζω ότι ο πρόεδρος ε, του Eurogroup ζήτησε μια εντολή για να μπορέσει να ξεκινήσει τις κατάλληλες επαφές. Νομίζω ότι τώρα θα έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος παρενέβη. Όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό στους συντονιστές, Υπήρξαν ε, πολλαπλέ απόψει σε σχέση με το ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα. Ένα θα μπορούσε να είναι ένα είδου συμφωνία ότι ε, θα ε, πρέπει να συζητηθεί το θέμα του διορισμού ε, ατόμων και από τα δύο φύλλα στα δικαιωτικά συμβούλια των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Και έτσι λοιπόν, ε, ίσω ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα χαρτί πορεία ε, για την ισότητα των δύο φύλων, για την συσσωροποιημένη εκπροσώπηση. Άλλοι πρότεινα να ξεκινήσει η διαδικασία με έναν άλλο διορισμό, αν και αυτό απερίφθη από τον πρόεδρο του Eurogroup, στη βάση ότι έχουν υλοποιήσει τις διαδικασίες μέχρι τώρα σύμφωνα με τα όσα λέει η συνθήκη. Νομίζω ότι τελικά αυτοί όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να αναλάβουν δράση απέναντί μας και ελπίζα ότι θα λάμβανα κάποια αντίδραση αυτή την εβδομάδα, αν όχι απευθεία τότε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά, όπως σας είπα, εγώ απλώς περιμένω να με ενημερώσουν. Δεν μπορώ λοιπόν να καθορίσω πότε θα γίνει η ακρόαση γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τέλματος και δεν μπορώ να πω καν στους συντονιστές ε, ορίστε αυτή την ενημέρωση είχα επίσημα μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε. Έχουμε την Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να επικεντρωθείτε για το αν αναρωτιέστε αν ε, θα καθορίσουμε ένα ραντεβού μέσα σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, γιατί τότε έχουμε την Ολομέλεια, είναι η τελική ψηφοφορία και ουσιαστικά είναι θέμα της Ολομέλειας. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω, αυτά γνωρίζω. Μάλιστα, σας ευχαριστώ και να προχωρήσουμε και θα τηρήσω τους συντονιστές και όλους τους υπόλοιπους ενημερωμένους ε, για όσα γνωρίζω. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Θεόδωρο. Νομίζω ότι μέχρι τις 11.30 θα προεδρεύσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να επιδιώξω κάποια άλλα ζητήματα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Πρέσ εδώ για την ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ε, Επιτροπή στη τέλη Μαΐου δημοσίευσε την έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Κάποιες μέρες αυτό το παρουσίασε ο κ. Σελμούνια σε αυτήν την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Και εγώ παρέδωσα το σχέδιο εκθεσής μου στις 17 Ιουλίου. Σήμερα θα κάνω την παρουσίαση της έκθεσης αυτής, της γνωμοδότησης αυτής και θα κάνω κάποιες προηγούμενες παρατηρήσεις. Καταρχήν, πρόκειται για μια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού που για πρώτη φορά υλοποιείται αφού έχουμε λάβει μια έκθεση όπου η Κομισιόν ζήτησε μια αλλαγή στη θεματική δομή. Μέχρι σήμερα η Κομισιόν ε, στην έκθεσή της παρουσίαζε τι κύριε τις κύριες πτυχές της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής αντιτράστ, ε, της πολιτικής κατάχρηση τη των κρατικών ενισχύσεων και έλεγχο των συγχωνεύσεων. Αυτά ήταν τα κύρια κεφάλαια που είχαν να κάνουν με τις ε, κύριες ερμοδιότητες, του κύριους τομείς της πολιτικής ανταγωνισμού. Τώρα αυτό αποτέλεσε τμήμα του εγγράφου εργασίας που εξαρτάται στην έκθεση. Η έκθεση ακολουθεί μια θεματική δομή για να τονίσει πως η πολιτική ανταγωνισμού συνεισφέρει στο να απαντήσει στις κυρίες προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δομή ε, είναι θετική κατά την άποψή μας γιατί απαντά στα αιτήματα της ομάδας ανταγωνισμού της Επιτροπής αυτής έχει διατυπώσει στην Κομισιόν τα τελευταία έτη. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση που για πρώτη φορά έχει μια θεματική δομή και που για πρώτη φορά αντικατοπτρίζει κάποια από τα κυρία ζητήματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο. Αυτό μπορούμε να σε επιτρέψει να εντοπίσουμε καλύτερα τους στόχους, ε, τις αρμοδιότητες ε, και τη συνεισφορά τους. Επίσης, ε, να σας πω ότι στην έκθεση προτείνεται η πολιτική του ανταγωνισμού. Όχι μόνο έχει το ΜΕΚ διάσταση, αλλά και θα είναι πολύ σημαντικό οι στόχοι της να επιδιωχθούν συνολικά στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να υπάρχει τέτοια παρουσία στο σύνολο των πρωτοβουλίων που παρουσιάζονται από την Κομισιόν στους διάφορους τομείς. Οι κύριε πτυχέ τη έκθεση αυτή καταρχήν έχουν να κάνουν μεταξύ τα εξή. Πώ απαντάει η πολιτική ανταγωνισμού στην κρίση, όταν βρισκόμαστε στο πέμπτο έτος ε, της ύφεση και ήδη θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια πιο συγκεκριμένη κρίση που έχει στο κέντρο της την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ακολουθώντας ε, και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην ομάδα εργασία, πώς δημιουργεί θέσεις εργασίας ε, και δημιουργεί ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη πτυχή έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, πώς διαρθρώνονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η τέταρτη πτυχή έχει να κάνει με το πώς προωθείται η ευημερία των καταναλωτών, και εδώ επικεντρωνόμαστε κυρίως ε, σε μια πολύ σημαντική παράγραφο που έχει να κάνει με τον ε, τομέα των τροφίμων ε, και ακολουθούμε μια σειρά σκέψεων για την αναγκαιότητα να υπάρξει νομιμότητα και αποτελεσματικότητα στην πολιτική ανταγωνισμού. Αυτές είναι οι κύριες πτυχές που προσεγγίζουμε στην παρούσα έκθεση. Τώρα, σε σχέση με την κρίση, υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με το αν η πολιτική ανταγωνισμού θα έπρεπε να βρίσκεται σε δευτερεύουσα θέση. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία των τελευταίων ετών ε, μας έδειξε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της πολιτικής ανταγωνισμού για να απαντήσουμε αποτελεσματικά στην κρίση. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι μία από τις ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και εκεί είδαμε ότι υπάρχει μια αποτελεσματική δράση όταν πρόκειται για αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων χρήσιμευσε για να προκαλέσει μεγαλύτερη σταθερότητα χρηματοοικονομική για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς και ταυτόχρονα είχαμε και πάρα πολύ ε, σημαντικές ε, ασφαλιστικές ε, ουσιαστικά ε, σε σχέση με την αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν προσπαθούμε να καθορίσουμε μηχανισμούς εξυγίασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν ο ανταγωνισμός ήταν πολύ χρήσιμος και επέτρεψε την καλύτερη χρήση των δημοσίων πόρων. Οι τράπεζες ε, που έχουν λάβει ένα είδους ε, κρατικής ενίσχυσης ε, και που λαμβάνουν άμεση ενίσχυση είναι προφανώς ότι πρέπει να μειώσουν το μέγεθός τους, να επικεντρωθούν ε, στο βιώσιμο επιχειρηματικό τους μοντέλους και να προσπαθήσουν να μειώσουν τον αντίκτυπο κυρίως ε, σε δύο μεγάλους τομείς, ε, τον αντίκτυπο έναντι των ανταγωνιστών που δεν έχουν λάβει ενισχύσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία και να έχουμε ε, ίσους κανόνες στον τομέα του ανταγωνισμού και να μειωθεί και ο αντίκτυπος επί των φορολογουμένων. Γιατί ουσιαστικά αυτοί ε, έχουν ε, τεθεί σε κίνδυνο. Έτσι λοιπόν προτείνεται να ακολουθήσουμε αυτές τις δύο σαφείς γραμμές στην πολιτική ανταγωνισμού. Όμως ε, οι δύο αυτές γραμμές θα είναι πάρα πολύ σημαντικές στο μέλλον για τις οντότητες που έχουν λάβει ενισχύσει ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εκεί ζητάμε η Κομισιόν ε, να ενισχύσει την πολιτική της για τον έλεγχο του ανταγωνισμού και τον έλεγχο των συγχωνεύσεων για να προωθήσει και να υπάρχει μια πιο ισορροπημένη συμπεριφορά. Και έτσι λοιπόν ε, λέμε στην Κομισιόν να συνεχίσει τις ερευνές της στην αγορά παραγόντων και ε, στο TC και στα CDS, τα credit default shops και επίσης στις υπηρεσίες πληρωμών όπως ε, και στι πληροφορίε που έχουν να κάνουν με τις χρηματαγορέ. Θεωρούμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να συνεχίσει να υλοποιεί έρευνα στους τομείς αυτούς και ήδη έχει ξεκινήσει την ανάληψη δράση ε, και επίσης ε, ζητάμε να παρακολουθεί τους πιο σημαντικούς, τις πιο σημαντικές εταιρείες και τον αντίκτυπο που έχουν στην αγορά. Επίσης γίνεται μια αναφορά ε, στα επεισόδια αστάθειας ε, των τιμών, στους οίκους αξιολόγησης και ζητάτε επίσης να συνεχίσει τη δράση της ε, σε ό,τι σε ό,τι αφορά την λειτουργία των επιτοκίων. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τους διάφορους δείκτες, το LIBOR, το EURIBOR, το DIBOR και θεωρούμε ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και τις ευθύνες του τομείς αυτούς σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό που τίθεται είναι ότι η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια ε, να έχουμε πιο εύρωστα δημόσια οικονομικά και συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωση για το 2020. επίση. το να έχουμε μια ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη, ε, κάτι τέτοιο στηρίζεται από την πολιτική ανταγωνισμού. Η ευφυή ανάπτυξη για να ε, τελειοποιήσουμε την εσωτερική αγορά και να πετύχουμε την ψηφική αγορά και για να έχουμε καινοτομία είναι προφανές ότι χρειάζεται ανταγωνισμός πολύ ισχυρό και φυσικά ανάπτυξη πάσας ευθύνη στο όλο το πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Ταυτόχρονα, σε ό,τι φορά στο περιβάλλον, πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις ε, τεχνολογίες που είναι πιο φιλικές για την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών μας στόχων ε, και τις κατηστητήριες γραμμές για τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακα, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τα σήματα που στέλνονται από τις τιμές και να μειώσουμε τις τρευλώσεις στην αγορά. Από την άλλη, ε, για ε, η πολιτική ανταγωνισμού προωθεί την πρόσβαση στην αγορά στα πλαίσια στρατηγική του 2020, πρόσβαση στην αγορά από την πλευρά όλων των πολιτών που υλοποιούν οικονομικέ δραστηριότητε ή που ε, έχουν επιχειρήσει. Η πολιτική ανταγωνισμού συνεισφέρει στην οικονομική πρόοδο και στο να διορθώσει τι ελλείψει τη αγορά και να υποστηρίξει τι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι η πολιτική ανταγωνισμού συνεισφέρει στην επίτευξη όλων των στόχων της στρατηγικής του 2020 και θα πρέπει ε, να την επιτελούμε σε ό,τι αφορά τι ε, Γενικέ υπηρεσίε, τι υπηρεσίε γενικού συμφέροντο, υπάρχει μια δεσμή μέτρων και ήδη το Κοινοβούλιο έχει πει ότι θέλουμε να υπάρχει μια πιο απλή μεταχείριση, μια πιο ευέλικτη μεταχείριση απέναντι στις υπηρεσίες αυτές με ένα πλαίσιο όπως υπηρεσίες, ε, όπως το χάρη τα νοσοκομεία, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές κατοικίες και οι υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος ε, κάτω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι θα πρέπει να εξαιρούνται από την φορολογία, να απαλλάσσονται θα πρέπει να απαλλάσσονται λοιπόν και θα πρέπει να δούμε τι έχει μεγαλύτερη σημασία από τι υπηρεσίε αυτέ σε αυτό το τομέα. Αυτό που μα ε, επισημαίνει την προσοχή είναι το τομέα των φαρμάκων και τη υγεία. Εκεί θα πρέπει να δοθεί σημαντική προσοχή, μεγάλη προσοχή από την πολιτική ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τα δικαιώματα ε, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ε, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής ε, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για τους πολίτες και είναι ένας τομέας σημαντικός στην οικονομία και έτσι λοιπόν η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αγορές και οι εμπορευόμενοι δραστηριοποιούνται σωστά. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, για τον καταναλωτή, εμεί επικεντρωθήκαμε στον τομέα του τροφίμων. Ο τομέα του να ε, έχει υψηλέ τιμέ τα τελευταία έτη. Υπάρχει αντίκτυπο λοιπόν ε, στι εγχώριε οικονομίε και στον πληθωρισμό. Το 14% του εισοδήματο των οικογενειών στην Ευρώπη δαπανάται στον τομέα αυτό έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή που τίθεται ένα νέο πλαίσιο και για τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις του τομείς αυτούς. Αυτό που επιθυμούμε είναι να διασφαλίσουμε ότι οι οργανώσεις παραγωγών θα ε, λειτουργήσουν ε, υπέρ του ανταγωνισμού και θα υπάρχει μια παρακολούθηση των τιμών των τροφίμων έτσι ώστε να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά. Επίσης, ξέρετε ότι οι διαφορές των τιμών δεν ε, ε, ωφελούσαν τελικά τους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει η πολιτική ανταγωνισμού ότι κατά μήκος όλης της αλυσίδας ε, λειτουργεί σωστά το σύστημα θα πρέπει τα δίκτυα ανταγωνισμού να διδικοποιήσουν το έργο τους σε αυτόν τον τομέα, κυρίως στα γαλακτοκομικά και στα παράγωγα προϊόντα, όπου είναι πολύ ευαίσθητα τα και το τελευταίο στοιχείο έχει να κάνει με την πρόθεση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής ανταγωνισμού. Δηλαδή, η νομιμότητα θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από το ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο αφενός, ε, θα πρέπει να υπάρχει μια λογοδοσία, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει έλεγχος της Κομισιόν, πάντοτε θα πρέπει να ακολουθεί τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι οι διαδικασίες στο πλαίσιο του ανταγωνισμού θα πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνεται για να διασφαλίζουμε πάντα τα δικαιώματα των πολιτών, κυρίως ε, τη δυνατότητα ε, να διατυπώσουν ε, κάποιες απαιτήσεις. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη και Ταυτόχρονα θα πρέπει να ευνοηθούν οι δυνατότητες ε, να θεσπιστούν ε, ε, κάποιες συμφωνίες έτσι ώστε να έχουμε ικανοποιητική έκβαση των διάφορων υποθέσεων για όλα τα μέρη. Θα πρέπει να ε, μην έχουμε αρνητικές συνέπειες ε, για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να μην υπάρχει αντίκτυπο στην απασχόληση. Όλε αυτέ οι τυχές θεωρούμε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίση, θέτουμε την αναγκαιότητα ότι ε, θα πρέπει να ελεγχθούν οι ευθύνε ε, των ε, επιχειρήσεων, όμως πέρα από αυτό θα πρέπει να απαιτήσουν και ανάληψη ευθυνών οι επιχειρήσεις από το προσωπικό τους. Η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να συμπληρώσει την αποτελεσματικότητα στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες εμπειρίες και να σκεφτούμε σχετικά με το θέμα αυτό. Επίσης, ταυτόχρονα υπάρχει αναγκαιότητα να συμπληρωθεί ο δημόσιος πυλώνας ε, με συλλογικές δράσεις και δράσεις από τον ιδιωτικό τομέα αποφεύγοντας ε, το σύστημα που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ή ε, να δημιουργούνται μη απαραίτητες διενέξεις. Και επίσης ζητείται από την Κομισιόν μια συνεργασία και στο πλαίσιο το με το ε, Ευρωπαϊκό Δίκτυο αλλά και με άλλους ε, τομείς για να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία κυρίως ε, σε αγορές που ένα είναι και πιο παγκοσμιοποιημένες και χρειάζεται όλο ένα και πιο πιο στην συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Επίσης αναφέρουμε και την ανάγκη περισσότερων πόρων για να έχουμε μια πιο προδραστική και αποτελεσματική πολιτική και επίσης απευθύνουμε έκκληση στην κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στο σχεδιασμό και στον έλεγχο των πολιτικών αυτών με ένα όλο ένα και πιο ενεργό τρόπο. Και εγώ θα θέλω να ευχαριστήσω τα διάφορα μέλη της ομάδας εργασίας ε, στο πλαίσιο του εγωνισμού για τη δουλειά που έκαναν και νομίζω ότι τους εκφράζω όλους όταν ε, ε, συγχαίρω και την επικεφαλής της γραμματείας. Ε, θα ήθελα να την ευχαριστήσω, αλλά και να την καλωσορίσω. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. We will start... ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσουμε με τους κοιόδης συγγητές, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να είστε όσο δυνατόν πιο σύντομο. Ο κύριος Γκίναρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση και το, η δουλειά του εισηγητή. Νομίζω πως ε, τώρα ο εισηγητής και ο προκατοχός του, Αντρέα Σφάμπ, πηγαίνουμε προς ε, ένα μέσο για να μετράμε την ζωτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, Μιλάω για την ετήσια έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί στην κρίση στην οποία είμαστε ε, μπορούμε πάντα να αναρωτιόμαστε αν έχουμε κάνει αρκετά όσον αφορά την εσωτερική αγορά και ελπίζω να συμφωνούμε όλοι ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά γιατί αν είχαμε κάνει αρκετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Και αυτό είναι μάλλον μία δυσάρεστη θεώρηση των πραγμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω δύο ακόμα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα η πτυχή των καταναλωτών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο ανταγωνισμός για τον καταναλωτή. Ο κύριος Πεσέδο τόνισε τον τομέα των τροφίμων. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω πως οτιδήποτε μπορούμε να πούμε για τα τρόφιμα, μπορούμε και πρέπει να το πούμε και για όλους τους υπόλοιπους τομείς της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Ακριβώς τα πράγματα εκείνα τα οποία επεσήμανε για τα τρόφιμα ο εισηγητής ισχύουν και για τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Το ζήτημα δεν είναι λοιπόν μόνο το 14% της ευρωπαϊκής οικονομίας φορά το 100% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Τίποτα λιγότερο. Και τίποτα περισσότερο. Βεβαίω πάνω από το 100% δεν γίνεται. Η άλλη ε, δε προοπτική είναι η δυναμική διάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε πως ο ανταγωνισμός δεν είναι ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων εταιριών. Ο ανταγωνισμός αφορά το να δώσουμε την δυνατότητα σε νέες εταιρείες, σε νέα προϊόντα και νέες προτιμήσεις και νέες ευκαιρίες. Και νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως αυτό το οποίο μας λείπει είναι οι νέες ιδέες, οι νέες εταιρείες, οι νέες δουλειές. Και, είπα αυτή την έννοια, θα έλεγα πως αυτή οι, αυτές οι αιτήσεις εκθέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να αναλάβουμε δράση σε αυτό τον τομέα. Νομίζω πως η Κομισιόν στο μέλλον θα επανέλθει σε αυτό το ζήτημα και ελπίζω να μπορέσουμε να εργαστούμε με βάση αυτή την ε, έκθεση. Δηλαδή να υπογραμμίσουμε πως εκεί όπου έχουμε ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός λειτουργεί, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι υγιής. Τα προβλήματά μας δεν βρίσκονται στους τομείς εκείνους όπου υπάρχει ανταγωνισμός. Τα προβλήματά μας κύριε Πρόεδρε είναι εκεί όπου δεν έχουμε ανταγωνισμό. Και δεν είναι αποδεκτό να δρανούμε. Γι' αυτό λέω πως θα πρέπει να έχουμε δύο προοπτικές και χαίρομαι που το συμπεριέλαβε αυτό στην εκθεσή του εισηγητής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τους κλάδους όπου υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού λόγω της νομοθεσίας. Αλλά είναι κυρίως λόγω της νομοθεσίας που συμβαίνει αυτό. Στο εθνικό επίπεδο και εκεί όπου δεν έχουμε μπορέσει να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες και άλλους τομείς. Και εγώ καλώς όρισα το ότι βεβαίως μπορούμε να συζητούμε τέτοια πράγματα ανοιχτά, αλλά πρέπει να δούμε και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Νομίζω πως ο δημόσιος τομέας και η ευθύνη του είναι να, να τα συμφέροντα των καταναλωτών, όχι των διαφόρων εταιριών, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, αλλά οι πάροχοι πρέπει να υποχρεώνονται να κάνουν ό,τι μπορούν για να δώσουν τις καλύτερες υπηρεσίες και αγαθά στους καταναλωτές και εκεί πέρα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Το δεύτερον, που πρέπει να τονίσουμε για να αυξηθεί η νομοποίηση αυτής της δουλειά και της έκθεσης είναι να τονίσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες πως εκεί όπου υπάρχει ανταγωνισμό είμαστε επιτυχεί. Και εκεί πέρα έχουμε τις νέες δουλειές και δεν θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας εάν δεν έχουμε ανταγωνισμό και ανταγωνιστικές εταιρείες σε διάφορους τομείς. Και, υπ' αυτή την έννοια κύριε Πρόεδρε, αναμένω την συνεργασία μου με τον εισηγητή για να αυξηθεί το επίπεδο των φιλοδοξιών του Κοινοβουλίου απέναντι σε Κομισιόν και Συμβούλιο και βεβαίως, όπως ανέφερε και ο εισηγητής, ένα κομμάτι το οποίο θα δούμε είναι οι κρατικές ενισχύσεις και πώς θα καταργηθούν σιγά σιγά για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να δούμε πώς μπορεί να αυξηθεί ο ανταγωνισμός σε όλους τους τομείς και στα τρόφιμα και σε άλλους τομείς. Νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα για να τονίσουμε τη σημασία που έχουν αυτά για τους Ευρωπαίους πολίτες, τονίζοντας τη σημασία του ανταγωνισμού. Όπως είπα, ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο μεταξύ υφιστάμενων εταιριών, είναι και για το άνοιγμα της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Και νομίζω η σημερινή έκθεση είναι μια καλή αρχή. Ευχαριστώ κυρία Σόφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Θα προτείνουμε κάποιες ε, τροπολογίες για να προσθέσουμε περισσότερο στο κείμενό σας παρά για να το αλλάξουμε, όμως θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα για την ε, κοινή γεωργική πολιτική και πολιτική αλληλείας, γιατί από ό,τι φαίνεται ο εισηγητής εδώ πέρα υπονοεί πως η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική αλληλείας ή ε, η μεταρρύθμισή τους δεν επαρκεί από τη σκοπιά του ανταγωνισμού. Ε, η Κομισιόν βεβαίω είναι συλλογικό σώμα Οπότε αναρωτιέμαι ποιες είναι οι συζητήσεις μεταξύ των ε, υπευθύνων για τον ανταγωνισμό και την αλληλεία και τη γεωργία φετέρου. Γιατί νομίζω και ο Γκούναρ Χεκμάρκ το ίδιο έλεγε. Για να εφαρμοστούν οι κανόνες του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς και στη γεωργία και την αλληλεία. Δεύτερον, και δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπει αυτό στην έκθεση, αλλά νομίζω πως τουλάχιστον πρέπει να γίνει μια αναφορά το ζήτημα του, της χειραγώγησης του Λάιμπορ και του Euribor και βεβαίως θα μάθουμε και περισσότερα ε, εντό του μηνό, αλλά θα ήθελα να μάθω κάποια πράγματα από την Κομισιόν για το τι έχει γίνει. Γιατί η Κομισιόν ανακοίνωσε πως θα δημιουργηθούν νέα μέσα για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο αλλά κάποιοι άλλοι θεωρούν πως η Κομισιόν ήδη είχε τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και θα ήθελα να γνωρίζω τι έχει κάνει η Κομισιόν και γιατί δεν παρενέβη νωρίτερα κατόπιν. Το επόμενο σημείο στην ειδική διάταξη αφορά τις κάρτες, τις πληρωμές, ε, ζήτημα των και βεβαίως δεν έχει ληφθεί καμία πρωτοβουλία. Ε, βεβαίω έχουν ε, καταλήξει υποθέσει στα δικαστήρια και αναρωτιέμαι γιατί η Κομισιόν αφήνει τα δικαστήρια να διαμορφώνουν την πολιτική αντί να αναλάβει η ίδια δράση. Και θα ήθελα να γνωρίζω το εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δράσει τώρα για να υπάρχει πραγματικά να, να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. Μας ενημέρωσε επίσης η Κομισιόν για το πολύ ανισχυτικό επίπεδο των αδικαιολόγητων κρατικών ενισχύσεων και δεν θυμάμαι ακριβώς τους αριθμούς, αλλά νόμιζα ότι ήταν γύρω στο 40%. Δηλαδή έπρεπε να χτυπάνε καμπανάκια. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες εξηγήσει. Τελευταία παρατήρηση για τις ε, συλλογικές πρόσφυγες. Εδώ πέρα νομίζω οι απόψεις θα διαφέρουν, θα αποκλίνουν εντός της Επιτροπής, ναι, πράγματι. Τουλάχιστον είμαστε συνεπείς ως προς την ασυμφωνία μας. Η Κομισιόν, από ό,τι φαίνεται, είναι αποφασισμένη να διατηρήσει κάποια αυτόματη εξαίρεση από τους γενικούς κανόνες διαφάνειας στο πλαίσιο της λεγόμενης ε, επιοίκειας. Κάποιες εξαιρέσεις μπορεί να δικαιολογούνται, αλλά αυτόματες εξαιρέσεις δεν νομίζω και νομίζω πως αυτός είναι ο κανόνας ε, όταν μιλάμε για διαφάνεια, πως κάθε εξαίρεση πρέπει να, δικαιολογούνται, να δικαιολογείται συγκεκριμένα. Και όσον αφορά τώρα την έκθεση Σάντσες εδώ πέρα, μια παρατήρηση που περισσότερο μπορεί να θεωρηθεί ηρωνική προστίκη. Λέτε στην παράγραφο, πως, ε, στην παράγραφο 3 πως το καθεστώς των ε, εκτάκτων κρατικών ενισχύσεων έχει διατηρήσει την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ε, είναι κάπως ειρωνικό γιατί δεν υπάρχει τέτοια σταθερότητα, αλλά για να σοβαρευτούμε στην παράγραφο 4 λέτε πως οι τράπεζε που λαμβάνουν κρατικέ ενισχύσει πρέπει να μειώσουν το μέγεθό του, να εστιάσουν το επιχειρηματικό του μοντέλο στο βιώσιμο τμήμα των δραστηριοτήτων του, να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπό του για του ανταγωνιστέ κτλ. Έχω τι αμφιβολίε μου για κάποια μέρη αυτής της ε, παραγράφου και είναι νομίζω πολύ χοντροκομμένος κανόνας για να ισχύσει σε κάθε ε, περίπτωση. Δεν πρέπει να γενικεύουμε νομίζω και γενικά να ζητήσουμε από τις τράπεζες να μειώσουν το μέγεθός τους. Οπότε προτείνω να σβήσουμε αυτή την παράγραφο. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να Είμαι συνοπτικός. Θα συνεχίσω σε αυτά που είπε ο Γκέναρ για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Είπε να εξασφαλίσουμε παροχή των κοινοφελών αυτών υπηρεσιών και να ασκήσουμε πίεση στους παρόχους για να το κάνουμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αν δούμε πώς λειτουργεί η αγορά και έχοντας γνώση για το θέμα αυτό, διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ κοντόφελμη η εστίαση σε άμεσο κέρδος, κάτι που δεν οδηγεί σε βιώσιμα συστήματα υγείας, παιδείας κτλ. Οπότε λέω με κάθε ειλικρίνεια ότι αν θα πρέπει να στηριχθούμε στις αγορές δεν νομίζω ότι θα εξασφαλίσουμε το μεγαλύτερο επίπεδο αποτελεσματικότητας υπό πιο μακροπρόθεσμη προοπτική γιατί δεν έχουν τέτοια προοπτική αγορές αν, είχα, αν ζούσαμε σε ένα ιδεώδη κόσμο, σε ένα ιδανικό κόσμο που θα δίνει μενάσματα στι αγορέ για την βιωσιμότητα, την κοινωνική, την περιβαλλοντική, ακόμη και την βιωσιμότητα του κέρδου, θα συμφωνούσα. Αλλά ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί έτσι η αγορά και παρά τι ατέλειε και, και την αναποτελεσματικότητα, ε, τα κράτη, οι κεντρικέ υπηρεσίε δεν είναι οι χειρότεροι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών. Σας έχω πει ότι για την υγεία τουλάχιστον ε, δαπανούμε το 11% του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Ε, στη, στις Ηνωμένες Πολιτείες 16% εμείς έχουμε πιο κρατικό σύστημα και με όλες τις μετρήσεις ε, οι δικές μας επιδόσεις είναι πολύ καλύτερες. Δηλαδή εξοπλίζουμε καλύτερα τα κονδύλια μας με τα κρατικά συστήματα που έχουμε εμείς τα δημόσια σε σχέση με τα ιδιωτικά που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πρέπει λοιπόν τυφλά να εμπιστευόμαστε τους ιδιώτες ε, ότι αυτοί θα κάνουν το καλό και ε, οι κρατικές αρχές κατά ανάγκη το χειρότερο. Σίγουρα η έκθεση αυτή δεν θα είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν μπορούμε να το φορτ να τη φορτώνουμε με απαιτήσει. Καταρχήν, ως προς τη δεύτερη γενική παρατήρηση, εκεί που λέει ότι οι συγκεκριτές θα πρέπει να λειτουργούν οι αγορές ικανοποιητικά για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα όμως ενδιαφερόμαστε για τους ε, πολίτες, ε, για τους ανθρώπους. Γιατί γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ καταναλωτών και πολιτών. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για φορολογούμενους, αλλά καλύτερα να λέμε για, για τους ανθρώπους. Και αν λέμε κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι εννοούμε πως οι αγορές θα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο που δεν θα παραβλάπτει τον πλανήτη, τη δυνατότητα του πολίτη να εξασφαλίσει ένα βιότοπο και υγιεινό περιβάλλον για τους ε, ανθρώπους. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο λείπει από την έκθεση και αυτή η παράληψη μας ανησυχεί. Θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες. Με στο 207. Είμαστε υπερβολικά μεγάλα ε, χρηματοπιστωτικά όργανα για να αποτύχουμε. Τώρα έχουμε ακόμη πιο μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα. Και αν αυτά δεν αποτελούν απειλή στην ε, εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τότε τι αποτελεί απειλή. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για το ζήτημα αυτό και πρέπει να κρίνω από τα αποτελέσματα το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με προβληματίζει ότι πόρο έχουμε ακόμη από το στόχο μας, δηλαδή τη μείωση, για να μην πω την εξάλληψη την, ε, της ίδιας έννοιας ε, των ε, too big to fail, παρά είναι μεγάλος για να αποτύχει. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοιες, τέτοια ιδρύματα, τέτοιους φορείς υπερβολικά ογκώδεις, γιατί από μόνοι τους αυτοί οι φορείς παραμορφώνουν την αγορά, έχουν τέτοια τεράστια ισχύ στην αγορά που εξορισμού την διαταράσσουν. Και επίση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όχι μόνο δυνατότητα ανταγωνισμού, αλλά και δυνατότητα νέων, νεοεισερχόμενων να μπουν στην αγορά και να είναι ανταγωνιστικοί. Το αντίθετο συμβαίνει. Ω προ την καινοτομία, όντω, είχαμε υπερβολική καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, το αντίθετο. Και αν καινοτομία σημαίνει ε, επαναφορά στον παλιό βαρετό τρόπο συγκέντρωσης ε, ε, καταθέσεων και επενδύσεων που έχουν πραγματική αξία. Αυτό μπορεί να είναι καινοτόμο, γιατί δεν νομίζω ότι απασχολεί πια το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Τέτοια είδου καινοτομία θα μα ενδιέφερε. Αλλά να δούμε πώ, βλέποντα τη διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού κλάδου, διαπιστώνουμε ότι ανταγωνιστικότητα δεν έχουμε. Έχουμε και σήμερα έμεσο, για να μην πω άμεσε άμεσες από τι κυβερνήσει. Και ε, αυτό ένας πράσινος που βλέπει πώς λειτουργεί η αγορά δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Αυτά και θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες για την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέρκιαν. Το μικρό μου είναι Ντέρκιαν. Το επίθετό μου είναι Έπινγκ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πρεσέντο, για το σχέδιο έκθεσης που ε, περιγράφει σημαντικές αλλαγές και γεγονότα που έλαβαν χώρα τελευταία χρόνια που ήταν αρκετά ταραχώδη. Θα υποβάλω αρκετές τροπολογίες. Ε, το έχω κάνει ήδη μάλιστα για μερικές και θα τις ε, αναλύσω σήμερα. Έχουμε καταρχήν την ανταπόκριση στην κρίση, την αντιμετώπιση της κρίσης. Με έκπληξη βλέπω ότι ο κύριος Πρεσέντο ε, στηρίζει την διεύρυνση των κρατικών ενισχύσεων, ενώ πέρσι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να σταματήσουν αυτά τα υποτίθεται προσωρινά μέτρα. Το 2009, όταν ήμουν συγγετής για την έκθεση του ανταγωνισμού, ήδη είχα εκφράσει τους φόβους ότι τα προσωρινά μέτρα δεν θα είναι και πολύ προσωρινά. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ανασταλεί. Επίσης έχει γίνει έργο της Ευρωπαϊκής, έχει γίνει έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Περιμένω το περιεχόμενο των νέων προτάσεων και να δω τι προτείνει για το μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί φαίνεται ότι αυτά τα σχέδια δεν περιλαμβάνουν το χρηματοπιστωτικό κλάδο, από την αρχή τους τουλάχιστον. Ο κύριος Μπαρόζο είπε να, να διατηρήσουμε το κατεπήγον καθεστώς για τις ε, τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Είπε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, ένα μηχανισμό πιο αποτελεσματικό για τις κρατικές ενισχύσεις και να αποφύγουμε τις στρεβλώσεις αγοράς που προκαλούν οι ενισχύσεις. Επίσης, διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο συγγετής στην παρούσα κρίση ως άλοθη, ως πρόσχημα για να τροποποιήσει τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού. Γιατί απότερο στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού είναι να άρει τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου όσο και σημαντική είναι η κοινωνική ένταξη και σωμάτωση, δεν εμπίπτει στη, στην πολιτική του ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό και όχι λιγότερο και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Χέκμαρκ. Ο ανταγωνισμός μας οδηγεί σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, κάτι που μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή λόγω του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας που έχουμε στην Ευρώπη. Πέραν της κρίσης Ευρωζώνης, ε, αυτό που μας ε, προβλημάτισε είναι η συγχώνευση πολλών περιφερειακών τραπεζών στην ε, Ισπανία σε μία τράπεζα, την Bankia, που μετατράπηκε σε γίγαντα στο too big to fail, υπερβολικά μεγάλο για να αποτύχει. Ποιο είναι ο ρόλος των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού, τι ρόλο διαδραμάτισε η Κομισιόν και οι αρμόδιε αρχέ ανταγωνισμού και τι είπαν για τη συγχώνευση αυτή, γιατί αυτή η συγχώνευση ήταν που έχει σημαντικές συνέπειες για το ευρώ και την ευρωζώνη. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που θα πρέπει να είναι ουδέτερος παίκτη στην όλη διαδικασία. Δεν με πείθει πρόταση ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μεγαλύτερο λόγο στις δραστηριότητες αυτές ε, της γενική διεύθυνση. Ε, γιατί είναι σημαντικό ο ρόλο γενική διεύθυνση στη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και προτιμώ να ενισχυθούν οι πόροι της γενικής αυτής διεύθυνσης με απόσπαση προσωπικού από άλλες γενικές διευθύνσεις που δεν έχουν τόσο κέρια σημασία, γιατί η πολιτική ανταγωνισμού βρίσκεται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βλέπω άλλο και οδησηγητή, οπότε catch the eye. Ο κύριος Βαπ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω στο catch the eye. Είμαι συντάκτης της ε, τοποθέτηση τη Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς φέτος και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Σάντσες Φρεσέδο για την πολύ ακριβή του έκθεση και θα ήθελα να παραμείνουν σε αυτή την ακρίβεια οι συνάδελφοι γιατί μην ξεχνάμε πως η έκθεση αυτή θα έχει ε, νόημα εάν εστιαστεί σε λίγα και καλά πράγματα το Κοινοβούλιο. Και υπ' αυτή τη μορφή νομίζω θα καταθέσει. Και Τροπολογίε για το ΕΛΚΟ, κύριο κύριος ε, Χέκμαρκ. Οπότε έχουμε για πολλωστή φορά αυτή την έκθεση. Νομίζω πω είναι πολύ πιο ε, ευανάγνωστη αυτή τη φορά η έκθεση τη Κομισιόν. Θετικό αυτό και χαίρομαι. Και τώρα για αυτά τα οποία είπε ο κύριο ε, Έπινγκ, αν υπόσχεται περισσότερο προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, νομίζω πως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε ακριβώς για την επιβολή του δικαίου ανταγωνισμού από τις δημόσιες ε, αρχές. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να σημαίνει πως η Κομισιόν να προσλαμβάνει ε, συνεχώς περισσότερα άτομα. Εάν θέλουμε να εφαρμόζεται σωστά το δίκαιο του ανταγωνισμού, πρέπει να έχει ε, επαρκές προσωπικό βεβαίως η Κομισιόν, γιατί Αλλιώς αναγκάζεται πράγματι να καταφεύγει σε ε, ιδιωτικές εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά και βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολη από το να την έκανε η Κομισιόν Εξοφίτσιο. Βεβαίως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις σχετικές ε, νομικές πρωτοβουλίες της ε, Κομισιόν, ειδικά φέτος για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και νομίζω πως το βάρος που έδωσε ο κύριος Άντης ατρόφιμα στα τρόφιμα είναι πολύ ενδιαφέρον και εδώ πέρα έχει δίκιο ο Γιούναρ Είναι ένας κλάδος από τους πολλούς για τους οποίους ε, θα πρέπει νομίζω να ε, εφαρμοστεί το δίκαιο του ανταγωνισμού. Επίσης, ε, βάρος δίνεται φέτος στις κρατικές ενισχύσεις και πρέπει να συζητήσουμε το εάν πραγματικά το να ανέβουν τα όρια, τα κατόφλια είναι πραγματικά μια σωστή κίνηση. Πράγματι δημιουργείται έτσι περισσότερη ευελιξία, αλλά από την άλλη πρέπει να είναι σαφές πως χρειάζεται επιγόντως μια εξυγίανση των προϋπολογισμών σε όλα τα κράτη-μέλη και άλλα, άρα δεν νομίζω πως ε, είναι σωστό να ανεβάζουμε τα όρια, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση των ε, σχετικών πολιτικών. Και δεν νομίζω πως πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα η πολιτική ανταγωνισμού. Έχει πάρα πολλά σωστά σημεία ο κύριος Σάντσες ε, Πρεσέδο και στο σημείο 4 που ασκούν ε, κριτικοί φιλελεύθεροι συνάδελφοι. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο επικριτικός. Γιατί λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις οι τράπεζες, γιατί έλαβε κρατική ενίσχυση η τράπεζα μπάνκια. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ε, δεν μπορούμε να κρίνουμε όλα με το ίδιο μέτρο. Ε, οπότε θα πρέπει να βρούμε ακριβώς ε, την τομή μεταξύ κράτους και τραπεζών όσον αφορά την αφακελοποίηση των τραπεζών. Εδώ πέρα έχω τις αμφιβολίες μου. Αυτό το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι το σημείο 19 όπου λέει συγκεκριμένα η έκθεση πως είναι σημαντικά τα προγράμματα εσωτερικής συμμόρφωσης ε, και αναφέρεται επίσης συγκεκριμένα στην έκθεση στο σημείο 22 πως ε, χρειάζεται περισσότερους πόρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πως εδώ πέρα μπορούμε να συμφωνήσουμε διακομματικά και θα έλεγα πως ε, κάτι το οποίο θα έλεγε συνήθως η κυρία Ινετφέλντ σήμερα το παρέλειψε το σημείο 16 υποστηρίζει ενεργότερο ρόλο του Κοινοβουλίου. Νομίζω πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό ως Κοινοβούλιο κατεπηγόντος. Νομίζω λοιπόν πως η έκθεση του συναδέλφου Σαντσπερσέδο είναι μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για φέτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σάντσες Πρεσέντο και να μιλήσω για τον αγροεπιστηστικό τομέα και τα τρόφιμα. Είναι ένα θέμα που άπτεται άμεσα της κοινή γεωργικής πολιτικής και της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Φυσικά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει η πολιτική αυτή, οι δύο πολιτικές, στην ε, γενικότερη πολιτική του ανταγωνισμού. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα αυτές οι πολιτικές ε, διαχωρίζονται πλήρως από την πολιτική ανταγωνισμού. Η κοινή γεωρική πολιτική, δηλαδή η κοινή ελευτική πολιτική, αποδεσμεύονται πλήρως από την πολιτική ανταγωνισμού. Ενώ Πρόκειται για δύο πολιτικές ε, που απορροφούν ένα μεγάλο τμήμα των κοινών μας πόρων και θα πρέπει και αυτές να εφαρμόζουν ε, τον ισότιμο ανταγωνισμό. Ε, η Επιτροπή μας είπε ότι στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολιτική πραγματικότητα, σαν να ήταν αυτή άσχετη από την πολιτική της ανταγωνιστικότητας, του ανταγωνισμού. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξηγήσουμε με πολύ διαφανή τρόπο στη συζήτηση για την πολιτική του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ε, προβλέπεται διαδικασία διαβούλευσης και θα έχουμε και σεμινάριο για το θέμα αυτό στις 25 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αν θέλει φυσικά, και μετά θα επανέλθουμε στον εισηγητή. Παρακαλώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον εισηγητή μας να είναι όσο πιο λακωνικοί γίνονται. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστώ. Ε, καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεση του κ. Πρεσέντο ε, που λαμβάνει υπόψη πολλά από τα σχόλια και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ θετικός ο τόνος ε, και υποστηρίζει τις περσινές δράσεις αλλά και αυτές που εξακολουθούν να, να δρομολογούνται. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια γενική υποστήριξη τη, της νέας μορφής που θα έχει αιτήσει η έκθεση ανταγωνισμού. Θεωρούμε ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι τμήμα της απάντησης και της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομική ανάκαμψη και μάλιστα εφαρμοστικέ δράσεις στην πολιτική ανταγωνισμού στόχο έχουν την υλοποίηση των στόχων της εσωτερικής αγοράς και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού υποστηρίζει και άλλες πρωτοβουλίες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λαμβάνουμε υπόψη και τα άριθμα σχόλια που διατυπώθηκαν σήμερα. Θα τα λάβουμε υπόψη. Ε, θα επικεντρωθώ εδώ σε ορισμένα μόνο σημεία. Διαπιστώνουμε ότι συνεχίζει η αμέριστη υποστήριξή σας προς τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, προσφυγές κατά του Τραστ και θα συνεχίσουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για προσφυγές ε, για αποζημιώσεις σε περίπτωση παραβίασης ε, της νομοθεσίας κατά τον Τραστ. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, χαιρόμαστε που αναφέρεστε στην έκθεση ECN για τον τομέα των τροφίμων που δημοσιεύθηκε το Μάιο μετά από έτοιμα μάλιστα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητήθηκε να είναι πιο ανταγωνιστικές οι οργανώσεις των παραγωγών. Βέβαια, η γεωργία ως κλάδος θα πρέπει ε, να υποβάλλεται και αυτό στους κανόνες του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τα καρτέλ, διαπιστώνουμε ότι υποστηρίζετε και εσείς ε, τις ε, δράσεις μας και την σύσταση να χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διακανονισμού. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του 19 θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Το σύστημα εφαρμογής Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διοικητικό και στόχο έχει τις επιχειρήσεις, από προς επιχειρήσεις και όχι στους α, ιδιώτες. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή κυρίως προστήμων τέτοιου είδους κυρώσεων στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως να δούμε τι γίνεται σε περίπτωση που υπάλληλοι συμμετείχαν σε τέτοιες παραβάσεις. Είναι μια παράλληλη διαδικασία κυρώσεων για να αποτραπεί τέτοια εμπλοκή. Βέβαια το ε, μοντέλο που έχουμε δεν εμποδίζει η ανάληψη τέτοιων δράσεων και κατά προσώπων. Επίσης σημειώνουμε ότι συζητήθηκε κατά πολύ το θέμα του αξιόπινου χαρακτήρα ορισμένων δράσεων, αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συνένεση. ό,τι αφορά τα καρτέλ, η εισαγωγή ποινικών κυρώσεων για τους ε, ιδιώτες ίσως είναι σημαντικός μηχανισμός για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ε, κυρώσεων ε, πέραν των προστήμων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, γιατί πραγματικά τα καρτέλ μπορούν να είναι επιβλαβή και για τους ιδιώτες. Πάντως, οι πρόσφατες εμπειρίες που είχαμε στα κράτη-μέλη δείχνει ότι η ποινικοποίηση μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν η σχετική νομοθεσία, η ποινική νομοθεσία δηλαδή, εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να πληρούνται διάφορα κριτήρια. Ανάγκη ε, κατάλληλης ανάκρισης, έρευνας, ε, σωστή απονομή δικαιοσύνης και προθυμία των δικαστών να εφαρμόζουν τέτοιες ε, ε και ποινικέ κυρώσεις. Και πολλές χώρες όπως η Σουηδία και, τα, και οι κάτω χώρες εξέτασαν την πιθανότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων και τελικά μετά από μεστή και περιστατωμένη ανάλυση απέρριψαν αυτή την πιθανότητα. Βέβαια, ο εισηγητή ζήτησε μια σχετική ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η ανακοίνωση είναι το κατάλληλο εργαλείο για να ανταποκριθεί σε, στην ανάγκη καλύτερη ενημέρωση για το θέμα αυτό. Προτιμούμε να συνεχίσουμε το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσω αυτού να ενημερώνουμε είτε προφορικά είτε γραπτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε μέσω δημοσιορακράσεων και σεμιναρίων. Τέλος, ε, ακριβώς επειδή έχουμε πενιχρούς πόρους αυτή τη στιγμή, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την έκκληση του εισηγητού να εξασφαλιστούν απαραίτητοι πόροι στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένουμε την εξέταση και των τροπολογιών. Ευχαριστώ κύριος Πρεσέντο και παρακαλώ χρόνου φίδου. Ευχαριστώ. Για να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Είχαμε και κάποιους ε, από τους συζητητές ε, στις εκθέσεις που θετήσαμε τα τελευταία χρόνια, κυρίως τον πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας, τον κύριο Σάπα και τους ευχαριστώ για την εμπειρία τους και για τη γνώση τους. Νομίζω ότι θα συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό αυτής της έκθεσης. Μάλιστα, είχε γίνει μία πρόταση εισαγωγική για να δώσουμε ε, ζωή στη συζήτηση και στη συζήτηση ε, ήθελα να θέσω κάποιες από τις ανησυχίες, δεν ήθελα να έχω πολεμικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι οι κύριοι άξονες ε, των θεματικών ε, που προσεγγίζουμε είναι εδώ, η κρίση, πώς συνεισφέρει ε, η στρατηγική Ευρώπη 2020, αυτή η ανάπτυξη που πρέπει να είναι ευφυής και βιώσιμη και φυσικά η πολιτική ανταγωνισμού δεν έχει ως μόνο στόχο τη συμπερίληψη, αλλά ουσιαστικά μπορεί να συνεισφέρει εκεί η πολιτική ανταγωνισμού εδώ ε, ουσιαστικά το να μπουν ε, νέοι παίκτε στην εσωτερική αγορά είναι κάτι σημαντικό. Εμείς αυτό θέλουμε οι δημόσιες αρχές να έχουν ε, επαρκείς πόρους που να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ε, και ουσιαστικά κάποιες ε, κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιούνται για να παρασχεθούν ε, κάποιες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος τους πολίτες. Έτσι λοιπόν η πολιτική ανταγωνισμού έμεσα ή άμεσα μπορεί να, συνεισφέρει στην κοινωνική ολοκλήρωση. Δεν θέλουμε εδώ να αντιπαρατάξουμε την πολιτική ανταγωνισμού με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος γιατί Ουσιαστικά δεν θέλουμε να κάνουμε τη συζήτηση για το αν είναι συμβατός ο ανταγωνισμός ή όχι με μια ε, πολιτική υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, ε, ανεξάρτητα από την ιδιωτικοποίηση ή όχι των δημοσίων υπηρεσιών. Ε, αυτή είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερη αξία στις ε, δημόσιες υπηρεσίες, πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πολίτες μας με λίγους πόρους. Και η πολιτική διαδικονισμού μπορεί να συνεισφέρει πράγματι στην επίτευξη αυτών των στόχων. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κάποια στοιχεία ισορροπίας ε, στη συζήτηση αυτή, στοιχεία που θα είναι όλοι σύμφωνοι. Πρόεδρε, Νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίε τι οποίε αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλέ πτυχέ που μπορούν να διορθωθούν και να συμπληρωθούν και εγώ νομίζω ότι η δική μου αποστολή είναι να ακούσω ε, γενικά τη θέλει Επιτροπή και να ψάξω να βρω μια κατεύθυνση όπου όλοι θα συμφωνούν. Και εγώ νομίζω ότι βάσει της εμπειρίας που έχουμε είμαι αισιόδοξο και θα τα καταφέρουμε τελικά. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι η κυρία Ινφελτ θέλει κάτι να προσθέσει, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη από τον Σύλλητο. Ζήτησα το λόγο πριν να, να πάρει το λόγο, αλλά δεν με είδατε. Αναρωτιέμαι πώς διαρθρώνονται αυτές τις συζητήσεις. Ε, θέτουμε ερωτήσεις ε, στην Επιτροπή, αλλά δεν ε, λαμβάνουμε απαντήσεις. Εγώ έχω θέσει πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις στην Κομισιόν και δεν λάβαμε απάντηση. Με ρώτησα για τις πολυμερείς τραπεζικές προμήθειες, την υπόθεση στο δικαστήριο για το Λίμπορ και το Γιούριμπορ και δεν έλαβα καμία απάντηση. Ρώτησα τι, ποια είναι η θέση του σώματος της Κομισιόν, ε, τι γίνεται και θέλω να λάβω μία απάντηση σε αυτές ε, τις ερωτήσεις. Είπε η Κομισιόν ότι θα απαντήσει αργότερα. Θα ζητήσω από την Κομισιόν να στείλει απάντηση σχετικά με τα σχόλια που ακούστηκαν εδώ. Παρακαλώ, εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τα συστήματα πληρωμών. Έχουμε το σημείο αυτό να ακολουθεί στην ημερική διάταξη και αφορά αυτό το θέμα και έχουμε συναδέλφους εδώ που θα μπορούσαν να, ε, να σας ενημερώσουν περισσότερο σχετικά. Σε ό,τι αφορά τις ε, συνεχιζόμενες ε, έρευνες, ξέρετε ότι πολύ καλά ότι δεν είμαστε σε θέση να το σχολιάσουμε. Μάλιστα, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 4 Οκτωβρίου, εξέταση τροπολογιών 5 Νοεμβρίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ τον Ιανουάριο του 2013. Τώρα, ας περάσουμε στην έκθεση του κ. Σαμποτέρχο προς μια ενωπημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα μέσω του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων. Εδώ θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, σκεώδεις συζητητές με τους οποίους είχα μια πολύ καλή συζήτηση σήμερα το πρωί και για την πολύ καλή συνεργασία και φυσικά τη γραμματεία εικόνα ε, για τη βοήθειά της. Λοιπόν, ε, είχαμε 155 τροπολογίες που έχω λάβει, οι οποίες συμπληρώνουν και διευκρινίζουν την έκθεση που το σχέδιο εκθέσει που έχω προετοιμάσει και συμφωνώ με πολλέ από τι απόψει που παρουσιάστηκαν από του Οι περισσότερε αλλαγέ ε, στο σχέδιο κειμένου έχουν να κάνουν με τροπολογίες που έχουν να κάνουν ε, με ε, ουσιαστικά τις πολλές διατραπεζικές προμήθειες. Τα ΜΥΦ. Πιστεύω ότι με τις τροπολογίες το κείμενο θα γίνει πολύ πιο αυστηρό από ό,τι ήταν αρχικά. Όμως η ίδια η Επιτροπή θα αποφασίσει αν θέλει να προωθήσει ευρωπαϊκή απαγόρευση όλων των ΜΥΦ ή αν θα ενθαρρύνει την σταδιακή μείωση αυτών των προμηθειών. Εκεί που φαίνεται όλοι να συμφωνούμε είναι ότι τουλάχιστον ε, θα πρέπει τα ΜΥΦ να βασίζονται στο πραγματικό κόστος και να είναι πιο διαφανή. Και αυτή η ε, σαφήνεια χρειάζεται, η νομική σαφήνεια, αλλά η πλήρης κατάργηση των πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών επίσης ε, προτάθηκε. Έχουμε λοιπόν ε, κάπως ε, αντιφατικούς συμβιβασμούς ε, επιτάπητος. Βέβαια στη συνάντηση των σχεδόν συγητών ομόφωνα αποφασιστήκε ότι στην παράγραφο 10 του κειμένου πρέπει να ζητήσουμε το κείμενο που ζητά από την Κομισιόν μελέτη αντικτύπου σε σχέση με την απαγόρευση των ΜΥΦ. Και θα θέλαμε αυτή τη μελέτη αντικτύπου να τη δούμε το συντομότερο στα τέλη του έτους, αν είναι δυνατόν. Τώρα, ένα άλλο θέμα που τέθηκε στη συνάντηση των σκιωδών ήταν οι επιβαρύνσεις. Αυτό είναι ένα τομέα όπου έχουμε αποκλίνουσε απόψει επίση από την πλήρη απαγόρευση στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι την απαγόρευση των υπερβολικών επιβαρύνσεων ή μια νέα μέθοδο υπολογισμού για το κατάλληλο επίπεδο των επιβαρύνσεων. Στο θέμα αυτό, επίσης, Στη συνάντηση των συγκεντρώσεων συγητών αποφασίστηκε ότι θα ήταν σοφό πριν ε, λάβουν ε, τελικές αποφάσεις οι πολιτικές ομάδες ε, και να προχωρήσουν προς την απαγόρευση, ότι θα πρέπει να έχουμε μία μελέτη αντικτύπου για την επιβάρυνση και την απαγόρευση των επιβάρυνσεων. Την επιβαρύνσεων. Μία τέτοια μελέτη αντικτύπου από την Κομισιόν. Τώρα, Χαίρομαι που βλέπω ότι έχουμε σύγκληση απόψεων σε άλλα θέματα σημαντικά, όπως είναι η ασφάλεια προστασία των καταναλωτών και η πρόσβαση τρίτων στις πληροφορίες ε, των ε, τραπεζικών λογαριασμών και στο υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών. Άρχισαμε ήδη να βρίσκουμε κάποιους καλούς μεταξύ των ε, σκηγωδών συγητών και είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας. Τώρα, ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις των μελών της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεγητά. Η κυρία που είναι η πρώτη σκιώδη συγγήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπως ε, είπε ήδη ο εισηγητής, οι ομάδες έχουν παρόμοιες ιδέες όσον αφορά την τυποποίηση, διασυνοριακές τυποποίησεις ε, ε, την ε, σήμανση και την πρόσβαση τρίτων μερών στους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς επίσης και την ε, εκπροσώπηση όλων των διαφορεμένων όσον αφορά τις διοικητικές δομές για την, ε, τις δομές ασφαλείας τέτοιων συστημάτων πληρωμών και νομίζω πως θα μπορούσαμε να βρούμε συμβασμούς αλλά μετά όπως είπε ο κ. Στέρχο έχουμε και τις ε, χρεώσεις ε, και τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες και διάφορες τροπολογίες. Οι πολυμερείς τροπήθειες ε, ξέρουμε πως πάρα πολλές φορές είναι πολύ ψηλό σε σχέση με το κόστος που καλύπτουν, αλλά αντιλαμβανόμαστε πως τώρα αποτελούν τμήμα του επιχειρηματικού μοντέλου. Άρα, όπως είπε ο κύριος Στέρχο, χρειάζεται μια διαφάνεια στις προμήθειες και μια αξιολόγηση αντικτύπου από την Κομισιόν το συντομότερο δυνατόν για να δούμε τι ε, ρύθμιση χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά, οι επιπρόσθετες ε, χρεώσεις, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ε, δεν βασίζονται αυτές πάντα στο κόστος, ε, καμιά φορά είναι απλά για να προσθέτουν έσοδα. Και στην κατάσταση αυτή όσοι χρησιμοποιούν πιο ακριβές κάρτες ε, εποφελούνται καθώς έχουν το ίδιο επίπεδο πρόσθετων επιβαρύσεων και το κόστος πληρώνω όσοι χρησιμοποιούν πιο φτηνές κάρτες. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να τονίσω την τροπολογία με υπαριθμών 160 γιατί θα πρέπει νομίζω να γίνεται αποδεκτή μία κοινή μέθοδος ε, πληρωμών χωρίς ε, επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως παραδείγματο χάρη ηλεκτρονικές πληρωμές και βεβαίως δεν θα πρέπει ποτέ να ξεπερνάνε προς τις επιβαρύνσεις το κόστος ε, το άμεσο. Αυτό θα απαιτεί διαφάνεια του κόστους, διαφορετικά δεν θα μπορούμε να υπολογίσουμε το αποδεκτό επίπεδο πρόσθετων επιβαρύνσεων. Η ολική απαγόρευση ε, μπορεί να οδηγήσει σε κρυφό κόστος και να εξασθενήσει την θέση των μικρομεσαίων εμπόρων όταν προσπαθούν να καλύψουν το κόστος των πιο ακριβών καρτών. Οπότε τουλάχιστον ε, ως προς αυτό χρειάζεται μια αξιολόγηση αντικτύπου των πρόσθετων επιβαρύνσεων και πριν βγάλουμε κάποια τελικά συμπεράσματα μιλάμε για μια πράσινη βίβλο ακόμα αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα για το τι ε, θέλει το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Γι' αυτό χρειάζεται μια εξελόγηση που πριν πάμε στην ε, νομοθετική πρόταση της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριο Σπάντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Τέρχο, τον εισηγήτη εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο ε, με το πώς έχει κυλήσει η συζήτηση. Ε, μας, μας ανησυχεί και μας απασχολούν όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρονται εδώ πέρα, πολυμερείς διατραπεζικές ε, προμήθειες, πρόσθετες χρεώσεις, ε, αναμένω την άποψη της Κομισιόν. Ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει τι ακριβώς ε, πληρώνει. Εμείς αυτή την πορεία θα ακολουθήσουμε και νομίζω θα βρούμε ένα συμβασμό. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τους σκιοδησηγητές. Κυρία Σοφία Ινετφέλτ. Ευχαριστώ, θα είμαι εξαιρετικά λακωνική, γιατί καταρχήν όλοι είμαστε ευγνώμονε προ τον εισηγητή για την πολύ επικοδομητική του προσέγγιση και υπάρχει και μεγάλο βαθμό ε, σύγκληση για θέματα όπως η τυποποίηση, ε, διακυβέρνηση, πρόσβαση σε πληροφορίες για το λογαριασμό, co-badging, τα περισσότερα του ενός σήματα και όλοι συμφωνούμε ότι από τους βασικότερους στόχους ε, του εγχειρήματο αυτού είναι να ανοίξουμε τις αγορές και να επιτρέψουμε την καινοτομία. Σε ό,τι αφορά τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, MIFS ε, και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, surcharges, το θέμα είναι γιατί παρά τις επανειλημμένε εκκλήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αναλάβει ακόμη δράση και Τώρα φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου τα δικαστήρια θα αποφασίζουν για τι πολιτικέ μα. Ε, βέβαια χαίρομαι για την ομολογία τη σχετική του ΔΕΚ, τη τελευταία απόφαση, αλλά προτιμώ εμεί να χαράζουμε τι πολιτικέ μα και όχι το δικαστήριο. Τι δράση προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί οι πολυμερείς τραπεζικές προμήθειε είναι κάτι που συζητούμε ε, εδώ και πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι των προμηθειών αυτών ε, στην Επιτροπή μας αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ εύρωστες αυτές οι τραπεζικές προμήθειες, ούτε ή να ήταν, και είναι δύσκολο να τις απαγορεύσουμε να τις εξαλείψουμε Κάθε φορά αναβάλλεται για αργότερα αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε πια και σε έφθετο χρόνο. Βέβαια, Ίσως υπάρχουν κάποιες προφανείς αντιφάσεις μεταξύ των δύο συμβαστικών τροπολογιών που εξετάσαμε. Στην περίπτωση ε, της τροπολογίας για τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, οι αντιφάσεις είναι φαινομενικές, δεν είναι ουσιαστικές. Πάντως θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μελέτη επιπτώσεων το συντομότερο δυνατό και να μην περιμένει να εγκρίνουμε εμεί την έκθεσή μας για να ξεκινήσει τις εργασίες επί της μελέτης αυτής των επιπτώσεων. Σε ό,τι αφορά τις επιπρόσθετες ε, επιβαρύνσεις, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο ε, επιλογές. Θα πρέπει να διαλέξουμε ή θα τις ε, επιτρέψουμε τις πρόσθετες επιβαρύσεις ή θα τις απαγορεύσουμε ολοσχερός. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση για να δούμε ποια λύση θα επιλέξουμε και να μπορούμε να την ε, αιτιολογήσουμε και να την τεκμηριώσουμε φυσικά αυτή τη λύση. Γι' αυτό ε, συμφωνώ με την κοινή πρόταση των σχεδόν εισηγητών ε, να, γίνει, να συνταχθεί μελέτη επιπτώσεων και για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις. Δεν βλέπω τους άλλους δύο σκιώδεις εισηγητές. κυρία Σλή μια και ο κύριος Μπάθ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χουντή τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και από την έκθεση αλλά και από τη σημερινή παρουσίαση του εισηγητή μας ε, σχετικά με το πώς βλέπει τις τροπολογίες φαίνεται ότι σε αρκετά πράγματα συμπίπτουν οι απόψεις μας και αισθάνομαι μια ικανοποίηση ότι έχει τις ίδιες ανησυχίες με αρκετούς από εμά, τουλάχιστον και με μένα σε ορισμένα σημεία. Επομένως αυτό που θα ήθελα να πω στην προσπάθεια πράγματι το κείμενο να γίνει πιο συγκεκριμένο και πιο αυστηρό ε, θα έλεγα πρώτον ότι κατά τη γνώμη μου και κατά τη δική μας άποψη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προστασία των πολιτών και των καταναλωτών μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα με την έννοια η τάση να γίνονται οι πληρωμές με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σήμερα ή από μετρητά, με μετρητά δυστυχώς θα δημιουργήσει αν δεν πάρουμε υπόψη αυτή την πραγματικότητα δυσκολίες σε κοινωνικές ομάδες ή και σε πολίτες ή και σε πρόσωπα που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε υπόψη τουλάχιστον να τονιστεί στις τροπολογίες μας, ε, από τις τροπολογίες μας απορρέει αυτή η λογική. Κατά τα άλλα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω, βέβαια θα δούμε και την τελική διατύπωση, το πρώτο είναι ότι πρέπει οι ηλεκτρονικές ε, πληρωμές να είναι ασφαλείς, όσο ασφαλείς γίνονται με τα σημερινά δεδομένα. Είναι. Το δεύτερο ότι δεν πρέπει η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών να μετακυλιστεί όπως γίνεται σε βάρος των πολιτών και των καταναλωτών. Το τρίτο σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες που είναι υψηλέ έγινε μια συζήτηση. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να καταργηθούν αφού πάμε για ενωπημένο σύστημα. Και το τέταρτο σημείο και τελειώνω είναι ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστασία από περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης και από διαρροή προσωπικών δεδομένων. Με βάση αυτές τις σκέψεις έχουμε καταθέσει τροπολογίες. Ε, επαναλαμβάνω, μετέχουμε στην διαδικασία. Α, κατάλαβα ότι ο εισηγητής αρκετά από αυτά τα βλέπει. Ε, στην τελική διατύπωση να α, συμβάλλουμε ώστε να πλησιάσει τουλάχιστον σε αυτά που νομίζουμε ως προτεραιότητες σε αυτό το θέμα που μοιάζει τεχνικό αλλά δεν είναι καθόλου τεχνικό, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για την καθημερινότητα των πολιτών τουλάχιστον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και σε πολλά καλύφθηκα, θα επικεντρωθώ σε ένα σημείο να ευχαριστήσω φυσικά τον εισηγητή για την πολύ ισορροπημένη του έκθεση. Φαντάζομαι δεν θα καταπλήξω κανένα που θα ασχοληθώ με τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, γιατί ήμουν ε, εισηγητής ε, σε ένα παρόμοιο θέμα και όπως είπε και η κυρία Ίνδελ δεν καταφέρουμε να σκοτώσουμε αυτό το ιό. Δεν θέλουμε να το σκοτώσουμε, γιατί οι διατραπεζικές προμήθειες ε, δεν είναι κοινοφελής υπηρεσία. Είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιούν ορισμένα ιδρύματα και μάλιστα στην, ε, στις πληρωμή έχουμε διευρύνει και το πεδίο εφαρμογή και θα πρέπει να αμείβονται αυτέ οι δραστηριότητε. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τι διατραπεζικές προμήθειε όντω στο παρελθόν έγιναν κάποιε καταχρήσει. συμφωνώ, να τι αναγνωρίσουμε. Αλλά αυτό που λέμε εδώ και χρόνια είναι ότι οι προμήθειες αυτές είναι δικαιολογημένες από τη στιγμή που είναι διαφανείς και τεκμηριώνονται οικονομικά δεν είναι το ίδιο να ζητούμε την κατάργησή τους. Μας λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μόνο έξι χώρες εφαρμόζουν τις διατραπεζικές προμήθειες. Αν είναι μόνο έξι χώρες σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμες αυτές οι προμήθειες. Αν τη λογική αυτή μιλήσουμε και για άλλα θέματα, θα κρίνουμε πολλά περίτα και άχρηστα, γιατί πολύ σπάνια έχουμε και τι 27 χώρε που να εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα. Γιατί λοιπόν μόνο 6 χώρε εφαρμόζουν το σύστημα αυτό και όχι οι υπόλοιπε. Για τι υπόλοιπε χώρε, η αμοιβή τη Υπηρεσία πληρωμών, ακόμη και με τι κάρτε, γίνεται με άλλο τρόπο. σε ορισμένες χώρες... Ε, ε, πληρώνει κανεί ε, το βιβλιάριο επιταγών. Δεν μα λέει κανεί ότι θα πρέπει να το καταργήσουμε. Το θέμα είναι ότι από τη μια έχουμε διαφάνεια και από την άλλη έχουμε αδιαφάνεια. Γιατί για ορισμένου ε, τρόπου πληρωμή ε, έχουμε επιβάρηση που επιβαρύνει άλλον τρόπο πληρωμή. Αν θεωρείται αυτό εξισορρόπηση και ισότητα των καταναλωτών, διαφωνώ. Σε ό,τι αφορά τι τραπεζικές προμήθειε. θυμάστε ότι και στην Ολομέλεια ο Επίτροπο μας είχε πει ότι αυτό που έχει αποφασιστεί δεν, ε, για τις άμεσες πληρωμές δεν ίσχυε εδώ ίσως. Ζητήσαμε μελέτη επιπτώσεων. Συμφωνώ. Αλλά θα πρέπει αυτή η μελέτη των επιπτώσεων να γίνει με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, όχι με στόχο να καταδείξουμε την ανάγκη κατάργηση των διατραπεζικών προμήθειών, αλλά να δούμε πόσο στοιχίζουν, αν είναι δικαιολογημένε και αν δεν υπάρξει αυτό ο τρόπο αμοιβή ε, για τους ε, παρόχου υπηρεσιών πληρωμή για τις κάρτες τη πιστοτική, τι τώρα θα υπάρξει. Γιατί θέλουμε να ευημερούν οι επιχειρήσεις, να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να είναι ανταγωνιστικές και απ' την άλλη να λέμε ότι το κέρδος είναι επονίδιστο να το κόψουμε. Εξαρτάται με ποιο τρόπο γίνεται γιατί βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πολλά και στο εμπόριο. Α γίνει λοιπόν μια μελέτη επιπτώσεων για τι τραπεζικέ προμήθειε, αλλά έντιμη και αμερόληπτη μελέτη επιπτώσεων, για να δούμε όλα τα επιμέρου στοιχεία και να δούμε τι εναλλακτική λίστα προτείνουμε για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση που καταργήσουμε τι διατραπεζικέ προμήθειε. Ευχαριστώ κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η τροπολογία υπαριθμών 30 του κυρίου Φόξ με βρίσκει σύμφωνο. Λέει ότι είναι πολύπλοκο και ίσως ε, θα ήταν δύσκολο να παρέμβουμε σε μια αγορά που λειτουργεί καλά. Συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε σόφρονες γενικά και νομίζω ότι αυτό προσπαθούσε να πει και ο κύριος Όμως ε, θα υποστήριζα και θα καταθέσω τροπολογία σχετικά μαζί με άλλου, ότι αυτή η αγορά δεν λειτουργεί καλά. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάτι. Τουλάχιστον μερικές φορές ε, βλέπουμε τι γίνεται στις ΗΠΑ ε, και αυτοί έχουν περιοριστική προσέγγιση εκεί και το κόστος ε, για τους καταναλωτές μειώθηκε σημαντικά και νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι, αλλά φυσικά χρειαζόμαστε μελέτη αντίκτυπου και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί Όμω η αγορά δεν ε, λειτουργεί και πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα, θα έλεγα εγώ. Ευχαριστώ κύριο Σέπινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρου ε, του κύριου Φόξ. Λυπάμαι που δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συζήτηση, αλλά ευχαριστεί τον κύριο Τέρκο για τη συνεχιζόμενη δουλειά του στην έκθεση αυτή. Ο κύριος Φόξ υποστηρίζει την προσέγγιση του εισηγητή και ε, οι τροπολογίε του θέλουν να βελτιώσουν και όχι να τροποποιήσουν το κείμενο. Μπορεί να υποστηρίξει το πρώτο συμβαστικέ ε, τροπολογίε ε, που έχουν κατατεθεί. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πληρωμέ στο διαδίκτυο με κάρτε και μέσω κινητών μέσων είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα, θα πρέπει να θέσουμε εμπόδιο στην καινοτομία μέσω τη υπερβολική ρύθμιση. Πρέπει να αναπτύξουμε καλύτερα το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και να δημιουργήσουμε θέσει εργασία στη διαδικασία. Η ρύθμιση δεν θα έπρεπε να θέτει εμπόδια στην καινοτομία όταν η αγορά είναι στη διαδικασία ανάπτυξη. Ο κύριο Φόξ συμφωνεί με τι τροπολογίε που υπογραμμίζουν την ανάγκη να δούμε πόσο πραγματικά κοστίζουν οι πληρώμε με μετρητά όταν ε, σκεφτόμαστε πόσο ακριβώς μας εξυπηρετούν οι πληρωμές ε, με κάρτα, μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων. Επίσης, τα συστήματα, τα και τα τετραμερή, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο για να έχουμε ίσους κανόνες για όλους, ενώ θα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές στο πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Σε ό,τι αφορά τα MIF, πολυμερικές τραπεζικέ προμήθειες, ο κύριος Φόξ ε, θα ήθελε μία συγκλήση προς τα κάτω που να αντικατοπτρίζει τα πραγματικά τέλη ε, δηλαδή το κόστος τη επεξεργασία των πληρωμών, καθώ δεν υπάρχει σήμερα ρεαλιστική εναλλακτική για τα MIF, ο στόχο δεν θα είναι να σε απαγορεύσουμε αυτές τις προμήθειες, αλλά ε, να ε, αποτρέψουμε τις υπερβολικά υπερβολικές προμήθειες. Ο κ. Φόξ δεν θεωρεί ότι πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο, καθώ αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερε προμήθειε σε χώρε όπου σήμερα είναι χαμηλέ. Ο κύριος Φόξ καλωσορίζει τα όρια στις επιβαρύνσεις ε, που επιφέρει η οδηγία προστασία του καταναλωτή, δικαιωμάτων του καταναλωτή, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και δεν θα πρέπει το κόστος να δημιουργεί ε, πρόσθετες, ε, πρόσθετα ε, το κομπάτζιν, τα πολλαπλά σήματα θα πρέπει να είναι ουσιαστικά κάτι που να προσφέρεται αλλά το να είναι υποχρεωτικά θα μπορούσε να έχει κινδύνους για την ασφάλεια και για τη συμβατική ελευθερία. Επίσης δεν θεωρεί ότι θα πρέπει οι άλλες τράπεζες να έχουν ε, πρόσβαση στον λογαριασμό του καταναλωτή πέρα από την επιβεβαίωση του ναι όχι για τη συναλλαγή. Επίσης, ε, ευχαριστούμε τον ε, κύριο Τέρχο και θα υποβάλει αυτά πριν από την ψηφοφορία της έκθεσης. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάποιε γενικέ παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα από τη σκοπιά της ιστορικής αγορα πριν δώσω τον λόγο στον συνάδελφο για τι πτυχέ του ανταγωνισμού και των πολυμερών προμηθειών. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, από όσο ακούσαμε και οι τροπολογίες που προτάθηκαν συμφωνούν με αυτά τα οποία είδαμε στη δημόσια διαβούλευση, ειδικά από την πλευρά των χρηστών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί οι Επιτροποί Μπαρνιέ και Αλμούνια ε, επανέλαβαν επανειλημμένως πως ο τελικός χρήστης των ε, μέσων αυτών είναι ο καταναλωτής, ο οποίος πρέπει να είναι στο κέντρο της ε, πολιτικής μας. Και νομίζω τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα είδαμε και στη δημόσια διαβούλευση, τυποποίηση διασυνοριακά τέλη, επιπρόσθετες χρεώσεις και πολυμερείς προμήθειες. Οπότε, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, να σας πω ότι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Νομίζω πως ε, τις επόμενες εβδομάδες ε, θα έχουμε ένα πρώτο προσανατολισμό, δηλαδή από τον τεράστιο τομέα που καλύπτει το ζήτημα. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα εκείνα που θεωρούμε πως ε, πρέπει να μας απασχολήσουν άμεσα και όπως ε, αναφέρει και η Πράσινη Βίβλος, συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις θα έρθουν του χρόνου το πρώτο εξάμεινο το 2013 και για να σας καθησυχάσω είμαστε στην τελευταία φάση της ανάλυσης αυτής κάπου γύρω στον Οκτώβριο θα κάνουμε μια πρώτη δήλωση. Έχει ξεκινήσει ήδη μια αξιολόγηση, οπότε οπωσδήποτε θα ακολουθήσουν μελλοντικέ νομοθετικές προτάσεις και ε, μελέτες αντικτύπου. Τώρα για αυτά τα οποία αναφέρθηκαν επί της ουσίας να ξεκινήσω από τις ε, πρόσθετες χρεώσεις, κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Εμείς θεωρούμε πως κομμάτι των προβλημάτων όσον αφορά τις υπερβολικές χρεώσεις αντιμετωπίστηκε με την οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών, αλλά είδαμε στη δημόσια διαβούλευση πως υπάρχουν κριτικές για το ότι είναι πολύ ανομοιογενές το περιβάλλον στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει επιλογή να επιτρέπεται, από τα κράτη-μέλη να απαγορεύεται η επιπλέον χρέωση, Η κατάσταση αυτή λοιπόν συχνά οδηγεί σε σύγχυση. Οπότε εξετάζουμε τρόπους να υπάρξει μεγαλύτερη ομοιογένεια στην αγορά. Και βεβαίως ε, τα έχουμε εξετάσει στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας υπηρεσιών πληρωμών που αναμένεται αρχές του επομένου έτους και έχουμε κάποιες ενδείξεις για το που θα πάμε στην κατεύθυνση των επιπρόσθετων χρεώσεων για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά τώρα τα τέλη, τα τραπεζικά, νομίζω πως θα δώσω λόγο συνάδελφο. Ευχαριστώ. Θα, δώσω... θα απαντήσω και στο ερώτημα της κυρία Σίνετφελντ που αφορούσε ακριβώς τα διατραπεζικά τέλη. Εκεί πέρα η κυρία Ινετφέλντ ε, είπε πως δεν είναι ικανοποιημένη για το ότι η Κομισιόν δεν είχε κάνει ε, κάτι νωρίτερα και μόνο τώρα προσπαθεί να βρει κάποιους ε, κανόνες. Εγώ διαφωνώ ότι δεν κάναμε τίποτα. Εμείς ε, ασχολούμαστε με αυτό το τομέα εδώ και πάνω από 20 χρόνια και το γεγονό πως το δικαστήριο του Λουξεμβούργου το Μάιο ε, έβγαλε μια απόφαση για τα διατραπεζικά τέλη ήταν ακριβώς συνέπεια του ότι η Κομισιόν είχε ευθύσει μια απόφαση σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Οπότε ήταν ακριβώς η δράση της Κομισιόν που οδήγησε στην απόφαση του δικαστηρίου Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα για το ότι το δικαστήριο το Μάιο συμφώνησε με την Κομισιόν σε όλα τα σημεία της προσέγγισής μας για, τα, ε, για τις συλλογικές αυτές διατραπεζικές προμήθειες. Βεβαίως αυτό ε, δεν σημαίνει πως ε, θα φύγει βεβαίως η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Υπάρχει υπόθεση κατά της ε, Mastercard και έχουμε ξεκινήσει και διαδικασίες κατά της ε, Visa για τον ίδιο λόγο ουσιαστικά με την υπόθεση του Μαΐου έχει υπάρξει λοιπόν μια δήλωση των ε, αντιρρήσεων μας τον Μάιο. Επίσης η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Αυτό μένει πως μπορεί να απαιτείται ένα ενιαίος κανονισμός που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς αυτό το ερώτημα ετέθη στην Πράσινη Βίβλο και εδώ πέρα χαιρόμαστε βεβαίω ε, για τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως είπε και ο συνάδελφός μου ελπίζουμε να μπορέσουμε να κοινώσουμε κάποια επόμενα βήματα τον Οκτώβριο. Είναι λοιπόν θεμητό το ερώτημα και το αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να τονίσω όμως, επειδή είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, πως ενώ ε, εξετάζουμε το ζήτημα, προφανώς συνεχίζει και η εφαρμογή της νομοθεσίας και με βάση την απόφαση του Μαΐου. Τα σχόλια τώρα όσον αφορά τα διατραπεζικά τέλη και την αναγκαιότητά τους και το ότι βεβαίως δεν υπάρχει τίποτα το δωρεάν, καμία υπηρεσία δεν είναι δωρεάν. Ε, εδώ πέρα πρέπει να ξεφύγουμε από μια σύγχυση. Υπάρχουν δύο τομείς με διατραπεζικές προμήθειες. Μιλάμε για συναλλαγές άμεσης χρέωσης σε έξι κράτη-μέλη ε, που είναι κάτι το διαφορετικό από αυτό το οποίο συζητάμε σε αυτή την πράσινη βίβλο που μιλάμε για κάρτες πληρωμών και μέσω κινητών και στο διαδίκτυο. Αυτά λοιπόν ε, χρεώνονται οπωσδήποτε στα περισσότερα εθνικά συστήματα και στο σύστημα της Mastercard και της Visa και βεβαίως αυτό το οποίο συζητάμε εδώ πέρα είναι πως ακριβώς διαφέρουν αυτά τα επίπεδα και αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς είναι πως έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούμε ακριβώς γιατί διαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα επίπεδα, γιατί τα τέλη παραδείγματο χάρη που χρεώνονται χωρίς να το ξέρω καταναλωτής στην Πολωνία είναι πέντε φορές υψηλότερα από το Βέλγιο. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για την εσωτερική αγορά, για την ολοκλήρωση της αγοράς και είναι ένα από τα ζητήματα που ετέθη σήμερα στην Αλλά κανείς δεν λέει πως πρέπει να παρέχονται δωρεάν οι υπηρεσίες. Το πρόβλημα με τις ε, διατραπεζικές ε, προμήθειες είναι πως δεν γνωρίζει ο καταναλωτής ότι ε, τις χρεώνεται και τον κατευθύνουν προς την πιο ακριβή υπηρεσία χωρίς να το ξέρει. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που θέτουμε στην Πράσινη Βίβλο. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο πάλι στον εισηγητή, τον κύριο Τέρχο. Και παρακαλώ να είστε και σύντομος. Okay. Thank you. Σας ευχαριστώ όλους για τα επικοδομητικά σας ε, σχόλια. Τώρα δεν θα προβώ σε περαιτέρω σύνοψη, αλλά θα αναφερθώ σε κάτι που κάποιοι μας υπερθύμησαν, ότι φυσικά το κάνουμε αυτό για να ωφελήσουμε τον καταναλωτή. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν ε, συζητούμε αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα και είμαι σίγουρος ότι ο στόχος όλων είναι αυτός. Σας ευχαριστώ και πάλι και θα προχωρήσουμε σχετικά γρήγορα την επόμενη εβδομάδα. Θα εργαστούμε επί αυτού του θέματος. Μάλιστα. 26 Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ και θα ε, ψηφιστεί και στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Τώρα να προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση, την έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ τροποποίηση της οδηγίας 2009. Για έχουμε εδώ την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να είναι στο δυνατόν πιο σύντομοι. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Να χαρεί και ο κύριος Μαν. Να γεια σας. η ΟΣΕΚΑ είναι οπωσδήποτε επιτυχημένες σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μιλάμε για 5,95 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι επενδεδημένα σε ΟΣΕΚΑ και είναι τεράστια επιτυχία γιατί υπάρχει ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο και άρα έχουμε ε, μια διαβεβαίωση για τους ε, καταναλωτές ε, και βεβαίως εκεί πέρα τοποθετούνται και στα τα μία και άλλες επενδύσεις έχουμε εδώ πέρα λοιπόν να βρούμε ταμεία και άλλες επενδύσεις. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία γιατί βεβαίως πρέπει να δούμε αυτόν τον τομέα και να το ρυθμίσουμε προς το συμφέρον του καταναλωτή και για να δημιουργηθεί και εμπιστοσύνη σε αυτό το επενδυτικό προϊόν και από την άλλη βεβαίω να υπάρχει ο κίνδυνος εάν πάμε πάρα πολύ μακριά τα τα, τα κονδύλια και τα προϊόντα αυτά να κινηθούν σε άλλους τομείς οι οποίοι είναι, θα είναι μετά λιγότερο ρυθμισμένοι. Οπότε η πρόταση της Κομισιόν ρυθμίζει κάποια πράγματα σε πέντε τομείς, κατ' ουσίαν δηλαδή. Πρώτα απ' όλα καλύτερε απαιτήσεις στις ε, τράπεζες ε, οι οποίες είναι θέματοφυλακέ και στην ευθύνη τους. Εκεί πέρα λοιπόν το θέμα είναι να λύσουμε τα διδάγματά μας από το σκάνδαλο Μάντοφ γιατί πάρα πολλοί Ευρωπαίοι έχασαν τα λεφτά τους και το θέμα είναι να φροντίσουμε ε, όταν ε, υπάρχουν ε, διαχειριστές ε, επενδύσεων και τράπεζες που δρούν ως θεματοφύλακες να είναι σίγουρος ο καταναλωτής πως δεν θα πληρώσει τη ζημιά για μια δομή την οποία δεν μπορούσε να ξέρει. Η ευθύνη λοιπόν την οποία προτείνει η Κομισιόν είναι σωστή. Τι συμβαίνει λοιπόν εάν δεν μπορεί όμως να ανταποκριθεί σε αυτή την αστική ευθύνη ο υπεύθυνο, όπως στην περίπτωση Μάντοφ. Γι' αυτό ήταν λοιπόν τόσο σημαντική αυτή η συμφωνία που επετύχαμε στην έκθεση Όλε για την προστασία των επενδυτών, δηλαδή και για τις ΟΣΕΚΑ, εάν δεν μπορεί να αποζημιώσει κάποιος ο οποίος έχει την ε, ευθύνη σε μια τράπεζα ή ένα αποθετήριο τίτλων ή όποιος είναι ο θεματοφύλακας. Εάν λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει αποζημίωση, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ε, πληρώσει τελικά. Δεν είναι δυνατόν ως απλός καταναλωτής να γνωρίζει κάποιος ε, όταν υπογράφει μια σύμβαση πως ε, υπάρχουν ε, κίνδυνοι με άλλους ε, συμβαλωμένους με τους οποίους ο ίδιος δεν έχει συμβληθεί. Οπότε δεν πρόκειται για ζήτημα ηθικού κινδύνου, νομίζω είναι λογική προστασία του καταναλωτή. Δεύτερον, στο, όσον αφορά το καθεστώς των αμοιβών και των αποζημιώσεων να κινηθούμε στο επίπεδο το οποίο υπάρχει ε, διεθνώς, ε, στον τομέα δηλαδή των λιγότερο ρυθμισμένων εναλλακτικών επενδύσεων. Εδώ πέρα όμως ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η άποψη των συναδέλφων, ειδικά εδώ θεωρώ πως πάρα πολλοί άνθρωποι σκέφτονται μήπως τα συστήματα αυτά αμοιβών είναι προς το ε, συμφέρον τους γιατί βεβαίως ε, λογική ανταμοιβή θα έπρεπε να είναι αυτή η οποία ανταμείβει το να είναι τα συμφέροντα του επενδυτή μαζί με του ε, διαχειριστή των κεφαλαίων και σε αντίστοιχη περίπτωση να έχει και αστική ευθύνη ο διαχειριστής. Πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή, όταν τα ταμεία και η ΟΣΕΚΑ κινητοποιούνται, ε, δραστηριοποιούνται στις ε, αγορές ε, να υπάρχει βεβαίως η ανάλογη ανταμοιβή του διαχειριστή αλλά βλέπουμε πως όταν τα πράγματα πάνε στραβά δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα εάν έχει πάει σε αρκετά μεγάλο βαθμό η διαφάνεια του κόστους το οποίο πληρώνει ο επένδυτης. Αν υπάρχει λοιπόν αρκετή διαφάνεια για το ποιο είναι το πραγματικό κόστος διαχείρισης ε, τέτοιων κονδυλίων και ιδιαιτέρως ε, αμφίβολο βρίσκω εδώ πέρα την πρακτική η οποία ακολουθείται και αφορά τα τέλη διατήρησης ε, λογαριασμού. Εδώ πέρα Εμποδίζεται λοιπόν ο ανταγωνισμός ε, για... και δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα επενδύσεις ο επενδυτής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποια κίνητρα ή να γίνει κάτι σε αυτόν τον τομέα. Επίσης ε, θετική είναι και η τρίτη παρέμβαση της Κομισιόν για μια, για μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση των κυρώσεων για να έχουμε αν όχι τις ίδιες τουλάχιστον συγκρίσιμες ε, κυρώσεις και εδώ πέρα προτείνεται μία ελάχιστη εναρμόνιση κάτι το οποίο χαιρετίζουμε. Τώρα, η ΟΣΕΚΑ 5 είναι ένα σχετικά περιορισμένο θέμα. Πολλά από τα μεγάλα ερωτήματα ήδη παραπέμπονται στο ΟΣΕΚΑ 6. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και πάρα πολλοί επενδυτές αλλά και ΜΚΟ και διάφορες ενώσεις οι οποίες συμμετέχουν σε αυτήν την διαβούλευση βλέπουν μια εξέλιξη η οποία ίσως δεν ήταν αυτή την οποία επιθυμούσαμε. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει στις ΟΣΕΚΑ δεν είναι αυτό το οποίο φανταζόμασταν. Δηλαδή η δημιουργικότητα σε αυτόν τον τομέα ξεπερνάει κατά πολύ ε, αυτό το οποίο θα έλεγα πως αντέχει η αγορά και δεν ξέρω αν ε, θα έπρεπε να αφήσουμε όπως λέγεται όλα τα λουλούδια να ανθίσουν εδώ πέρα ε, αναμένουμε την άποψη κομισιών. Είναι νομίζω ξεκάθαρο πως θα πρέπει οι ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε ρευστά προϊόντα και δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ της ε, λειτουργίας αυτών των ΟΣΕΚΑ και της τοποθέτησης ε, σε οικολογικά ή πιο κοινωνικά χρήσιμους ε, τομείς. Και ε, βεβαίως έχω ξεκινήσει συζητήσεις με την Κομισιόν για το πώς η Κομισιόν θα μπορέσει να προωθήσει τον τομέα των επενδύσεων των οικολογικών και των κοινωνικά υπεύθυνων. Και βεβαίως αναμένω την περαιτέρω συνεργασία. Αναμένω λοιπόν να ακούσω τι θα πούν τώρα οι συνάδελφοι και είμαι σίγουρος πως ε, θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία έτσι ώστε η αγορά των ΟΣΕΚΑ να εξακολουθεί να λειτουργεί λογικά προς όφελος των καταναλωτών και εντός και μετά την ε, κρίση. Αυτά και σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Πέντε σκιώδεις έχουμε παρόντες. Θέλουμε παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ο κύριος Τόμας Μάν ο πρώτος. Ευχαριστώ και εγώ θα μιλήσω γερμανικά όπως μόλις έκανε ο Σβέν. Ξέρετε πως η πολιτική πάντα τρέχει ε, λαχανιάζοντας πίσω από τις αγορές για να διορθώσει αυτά τα οποία έχουν πάει στραβά. Γι' αυτό είναι θετικό το ότι έχουμε την δυνατότητα να αντιδράσουμε με την ΟΣΕΚΑ 5 και για την ε, προστασία των ε, επενδυτών. Οι επενδυτές εδώ πέρα είναι μικρο αποταμιευτές, ε, έχουν λοιπόν, είναι ιδιώτες πελάτες, έχουν ανάγκη υψηλής προστασίας, αυτό είναι γεγονός και πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να υπάρξει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Εάν το καταφέρουμε αυτό θα Έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα και νομίζω πως η πρόταση της Κομισιόν είναι σωστή. Υπάρχει υψηλή προστασία των επενδυτών ενδιαφέρον. Είναι επίσης πως ε, βλέπουμε πως ε, και οι θεματοφύλακες ε, πρέπει να έχουν κάποια ευθύνη. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Και κάτι ακόμα θα έλεγα πρέπει να εμπλέκονται αυτοί οι οποίοι παίζουν τον ε, ρόλο θεματοφύλακα αλλά βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός ε, ανάμεσα σε αυτούς και τους ε, ΟΣΕΚΑ. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στον σημαντικό αυτό τομέα να έχουμε και κυρώσεις και να υπάρξει όπως υπόθηκε μια ελάχιστη εναρμόνιση. Πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα πολλά διαφορετικά κασόντα να ε, εναρμονιστούν. Κάποιοι ε, επενδυτές δεν γνώριζαν τις δυνατότητες που είχαν. Νομίζω λοιπόν σας στείλουμε εδώ πέρα ένα καλό μήνυμα. Οι διαβουλεύσεις θα ακολουθήσουν οπωσδήποτε θα είναι ενδιαφέρουσες και είμαι σίγουρος πως θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία. Στόχος μας και μας είναι ο ίδιος. Εδώ πέρα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, τους επενδυτές και νομίζω πως είναι σε καλύτερη θέση ε, τώρα από ότι τα τελευταία χρόνια με τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία πρέπει επιτέλους να τελειώσουν. Ευχαριστώ κυρία Μακάρθη. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για την παρουσίασή του, με την οποία συμφωνώ και με την προσέγγιση του γενικώ. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία να χρησιμοποιήσουμε την αναθεώρηση αυτή τη νομοθεσία για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Γιατί είχαμε περιπτώσεις ε, κατάχρησης των ΟΣΕΚΑ και έχουμε ευκαιρία να διορθώσουμε κάποιε αδυναμίες και αναφέρθηκε στην υπόθεση Μάντοφ και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις που είχε στην απώλεια εμπιστοσύνη των επενδυτών. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί περιμένουμε τις κατηδίαν να συναντήσουμε τον εισηγητή. Θα ασχοληθώ με πιο γενικά θέματα εδώ. Θέλουμε σαφή ενημέρωση για, την, για το δανεισμό των κινητών αξιών, τις πρακτικές ε, κέρδους, τους κινδύνους και να ξέρουμε ποια νομική οντότητα είναι σε τελική ανάλυση θεματοφύλακας, υπό την εποπτεία ποιου και πώς ισχύει ε, η αστική ευθύνη για τα στοιχεία του ενεργητικού. Είμαστε υπέρ ενός αυστηρότερου καθεστώτος ε, ευθύνης. Θέλουμε μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας για τον επενδυτή. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να είναι σαφής η αποκάλυψη στοιχείων για τους επενδυτές ή τουλάχιστον για κάποια στοιχεία του ενεργητικού. Νομίζω ότι εκεί θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την αμαθεσία, Επίσης, ετήσια πιστοποίηση της θεματοφυλακής του στοιχείου του ενεργητικού και να δούμε ε, ότι αυτή η θεματοφυλακή γίνεται στο όνομα του πελάτη. Βέβαια, φαντάζομαι κάποιοι συνάδελφοι θα επικαλεστούν το επιχείρημα ότι αυτό θα επιβαρύνει περαιτέρω τον κλάδο, γιατί πολύ συχνά για να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη του επενδυτή επιβαρύνουμε τις, τα διάφορα ιδρύματα και τους φορείς. Θα δούμε αν υπάρχει απόδειξη ότι η πιστοποίηση συνιστά ε, επιπλέον επιβάρηση να το εξετάσουμε. Νομίζω όμως ότι τα ωφέλη θα είναι τόσο μεγάλα για τους επενδυτές που αξίζει τον κόπο, γιατί θα έχουμε μια πραγματική ε, σαφή εικόνα του συνόλου του, του συνόλου του ενεργητικού. Πάντως θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, με τον εισηγητή και τους Σκιώδης. Εν γέννη πάντως συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητού που στόχο έχει την ε, αποκατάσταση εμπιστοσύνης των επενδυτών, την τροποποίηση κάποιων σημείων για να αντιμετωπιστούν οι καταχρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και οι απόλυτες εμπιστοσύνη που έχουν δημιουργήσει. Η κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχήν να αναφερθώ στη δήλωση οικονομικού συμφέροντος, γιατί συμμετέχω στο ε, Συμβούλιο ενός ε, Συμβούλιο Επενδυτών και μάλιστα εκπροσωπώ ε, τους ε, επενδυτές, κυρίως επενδυτές σε ΟΣΕΚΑ. Συμφωνώ ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αξιέπαινη και όπως είπαν και προλαλήσαντες είναι σημαντικό να προτάξουμε την ανάγκη προστασίας των επενδυτών απέναντι στις τράπεζες. Επίσης θα πρέπει να θεσπίσουμε τους κανόνες που χρειάζονται για την αποκατάσταση εμπιστοσύνη και από αυτή την άποψη συμφωνούμε με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, ως προς τις λεπτομέρειες ε, θα γίνει περαιτέρω συζήτηση. Πάντως θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πολύ καλό προπαρασκευαστικό έργο με τις προτάσεις της. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα αποδοχών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη φυσικά και τα συμφέροντα των επενδυτών και να δούμε τι ε, ενάβσματα θα δώσουμε για την προστασία των επενδυτών. Είναι αρκετά απλή η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρησιμοποιείται η ίδια αρχή με αυτή ε, ενό άλλου νομοθετικού κειμένου της, οδη... της τα Ιδρύματα ε, Εναλλακτικών Επενδύσεων. Θα πρέπει όμως ε, να δούμε τις ιδιαιτερότητες της νέας πρότασης και φυσικά πώς θα εφαρμόσουμε τις διάφορες διατάξεις. Εμείς οι φιλελεύθεροι δεν θέλουμε ε, παρεμβάσεις στα συστήματα αποδοχών, αλλά είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε. Επίσης, οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι παρόμοιες στις ε, χώρες μέλη γιατί με το ΣΕΚΑ 4 θεσπίσαμε ένα μηχανισμό για την ενίσχυση των διασυνοριακών συναλλαγών. Οπότε είναι λογικό όταν έχουμε διασυνοριακές δραστηριότητες και τα συστήματα κυρώσεων να είναι συγκρίσιμα με τι άλλο. Τώρα, κάποιες αντιρρήσεις που αναφέρθηκαν. Η κυρία Μακάρθη είπε ότι ο τραπεζικός ο, τομέ, ο τραπεζικός τομέας θα διαμαρτυρηθεί για τις απρόσθετες επιβαρύνσεις ε, λόγω της πιστοποίησης για παράδειγμα. Αλλά έχουμε και άλλα επιχείρηματα. Έχουμε τις ε, τράπεζες που είναι θεματοφύλακες, ε, είναι θεματοφύλακες για στοιχεία ενεργετικού τρίτων χωρών. Εκεί πέρα σε τέτοιες περιπτώσεις ποιος φέρει την ευθύνη. Νομίζω ότι το ζητούμενο εδώ είναι να φροντίσουμε εξασφάλιση των επενδυτών και εγγύηση ότι οι επενδύσεις τους θα τύχουν προστασίας. Ευχαριστώ, κύριο Κάμαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ε, τον συγχυτή και μάλιστα πριν από την υλοποίηση της συζήτηση αυτής είχαμε αρκετές συζητήσεις για τους ΟΣΕΚΑ και ξέρω ότι είχε συζητήσει με άλλους σκιώδεις ε, και με κάλεσε και σε μια εκδήλωση στο Λονδίνο και νομίζω ότι κάποιες από τις ιδέες που συζητήσαμε εκεί σε σχέση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογή των ΟΣΕΚΑ και σε σχέση με το ATF ε και τη δομή του ήταν ε, κάτι θετικό όμως εγώ νομίζω ότι στη νέα πρόταση της Κομισιόν του 2016 θα ήταν το κατάλληλο πλαίσιο να ρυθμιστούν αυτά ο λόγος που καλωσορίζω αυτή την πρόταση για τους 15 είναι γιατί όταν ε, εξετάζουμε διάφορα στοιχεία ε, βάση, ε, μάλλον και λόγω της οικονομικής κρίσης, διάφοροι αναφέρουν την υπόθεση Μάντοφ ε, και εκεί θεωρούσαν ότι αυτό ήταν ε, ουσιαστικά ένα ε, ταμείων βιών κεφαλαίων και ότι έπρεπε να έχουμε εκεί τους κατάλληλους κανόνες. Όμως εδώ και για τα αποθετήρια πρέπει να ρυθμίσουν κατάλληλους κανόνες και να έχουν κάποια ευθύνη. Δεδομένων των ε, ε, αλλαγών που κάναμε στην οδηγία για το διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, νομίζω ότι θα ήταν απαράδεκτο για τους γενικούς επενδυτές να έχουν λιγότερη προστασία από τους επαγγελματίες επενδυτές. Υπάρχουν ε, κάποιοι τομείς που θα ήθελα να διερευνήσω περαιτέρω. Ένας από αυτούς τους τομείς ε, θα είναι αν ε, μπορούν να απαλλαχθούν οι θεματοφύλακες από την ευθύνη, αν το απαιτεί αν η εθνική νομοθεσία απαιτεί να χρησιμοποιήσουν έναν υποθεματοφύλακα. Εγώ νομίζω ότι πολύ συμφωνούμε ότι τελικά θέλουμε κάποιον να είναι εν τέλει υπεύθυνο. Κάποιο πρέπει να έχει μια ευθύνη. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογία απλώ για να απαλλαχθεί από την ευθύνη. Αν δείτε στην κρίση, ε, σε όλο τη το φάσμα, νομίζω ότι αυτό που μα ενόχλησε όλου είναι ότι οι διευθυντέ των τραπεζών που δεν τα πηγαίναν καλά δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Θέλουμε όμω κάποιο να αναλαμβάνει ε, την ευθύνη για αυτή την επιτυχία στο όλο το χρηματοπιστωτικό τομέα. Διαφορετικά υποσκάπτει την εμπιστοσύνη μας. Επίση, αναρωτιέμαι για αυτή την απέτηση ο φίλακάς ε, να είναι ε, ρυθμιστή σε ένα πιστωτικό ίδρυμα είτε στο ΜΥΦΙΤΕ. Κάποιοι ε, τραπεζικοί μου είπαν ότι είναι παράλογο και πρέπει να το δούμε αυτό γιατί λένε κάποια ιδρύματα ότι θα αποκλείονταν χωρίς να χρειάζεται και δεν ε, ωφελεί κάτι τέτοιο τους επενδυτές. Ίσως δηλαδή μπορεί να οδηγούμε σε συγκέντρωση, σε συγχωνεύσεις αν ε, αφαιρούμε κάποιους προαράγοντες από την αγορά. Έτσι λοιπόν, ε, τότε θα έχουμε κάποια συγκέντρωση και μεγεθύνουμε τους κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να το διερευνήσουμε αυτό το θέμα στις συζητήσεις μας. Και στη μελέτη που έγινε κάποιος ε, λόγος ε, για το θέμα αυτό, μπορεί να φυγούν ε, και κάποιοι μεσάζοντες. Αν δούμε το θέμα των κυρώσεων, θα ήθελα να υπάρχει ευθυγράμμιση με την οδηγία, με τη διαφάνεια, δηλαδή να έχουν οι αρμόδιες αρχές ένα ρόλο να διαδραματίσουν. Νομίζω ότι αρχή θα πρέπει να είναι η διαφάνεια και νομίζω ότι συμφωνούμε στο ότι θέλουμε περισσότερη διαφάνεια για να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία, έτσι ώστε να λαμβάνουν οι επενδυτέ τι πληροφορίε που χρειάζονται, αλλά να μην του επιβαρύνουμε και υπερβολικά. Και τέλο, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ε, ε, ε, ε, ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα, δηλαδή ότι δεν υπήρχε ευθυγράμμιση μεταξύ των διάφορων συμβουλίων. Ε, σε σχέση με τις ε, επιδόσεις των επενδύσεων. Ε, κάποιος μίλησε για το ρόλο των εμπειρογνωμόνων ουσιαστικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσό τιμαριθμητικής προσαρμογής. Όταν λοιπόν οι εμπειρογνώμονε δεν τα πάνε καλά, δεν θα πρέπει να αποζημιώνονται για αυτέ τι κακέ επιδόσεις. Θα πρέπει η αμοιβή του να συνάδει με τι καλέ επιδόσει ή θα πρέπει με δείξουν να δούμε τι επιδόσει όπως και να έχει. κυρία Λούλινγκ, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πω, καταρχήν, ότι δεν υπάρχει κανείς εδώ που να μην υπογραμμίζει την αναγκαιότητα βελτίωση της προστασία ε, των επενδυτών ε, στο πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ. Θα ήθελα να κάνω καταρχήν μια παρατήρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα εργαζόμαστε για το ΣΕΚΑ και ήδη ανακοινώνεται και η πρόταση για τον ΣΕΚΑ 6. Εγώ αναρωτιέμαι μήπως θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια πιο πλήρη αναδιατύπωση της νομοθεσίας για τους ΣΕΚΑ. Σε λιγότερα τακτικά χρονικά διαστήματα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι σόφρον συνεχώς να τροποποιούμε την νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τη 5, για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές ε, στην νομοθεσία για τους οσέκα, με στόχο την εναρμόνιση των προτύπων ε, των θεματοφυλάκων ε, σε υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη το περιεχόμενο της ε, οδηγίας ε, IFM, διαχειριστής οργανισμών ελλακτικών επενδύσεων. Αυτή η οδηγία ε, εισάγει ένα ιδιαίτερα πλήρες νομικό πλαίσιο και τελικά λέει ο ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να ενισχυθούν από ένα σύνολο κανόνων. Έτσι, λοιπόν, ο κύριος στόχος θα έπρεπε να είναι μια σύγκληση των ε, προτύπων ε, μεταξύ του AFM και του ΣΕΚΑ5. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την ε, εποπτεία από την πλευρά των αρχών και θα επέτρεπε να έχουμε ίσους κανόνες για τη μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων και να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Και τελικά θα διευκολύναμε και τον τομέα ε, των επενδυτικών κεφαλαίων ή οσεκά ουσιαστικά έχουν σχεδιαστεί για τους επενδυτές σε ελληνικό επίπεδο, για τους μη επαγγελματίε και θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι η αρχή εποπτείας, ο θεματοφύλακας και ο διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ και η συνεργασία μεταξύ τους είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να πω ότι καταρχήν θα πρέπει να ε, εστιάσουμε σε μια σύγκληση με τους υψηλούς κανόνες, με τα υψηλά πρότυπα που προτείνονται από την οδηγία EFM. Δεύτερο, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ε, των οντοτήτων, προστατεύοντας τους επενδυτές και τρίτον να έχουμε μία σαφή κατανόηση του αντικτύπου του κανόνων ε, ανάθεσης σε ορισμένες αγορές και για ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού. Ξέρετε ότι ο διάβολος κρύβεται πάντα στις ε, λεπτομέρειες και εδώ μιλάμε για τεχνικές ε, λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την προστασία των επενδυτών. Και το σύνολο της ε, ε, δομής των ΟΣΕΚΑ, γιατί εμείς ε, ουσιαστικά θεωρούμε ότι ο ΟΣΕΚΑ είναι πραγματικά ευρωπαϊκή επιτυχία και μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τελικά η κυρία Λούλινγκ με κάλυψε πλήρως. Ήμουν ε, εισηγητής για τη ΣΟΣΕΚΑ το 2001-2003 και για 13 χρόνια κολλήσαμε και δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Ήταν ε, τεράστια η επιτυχία των ΟΣΕΚΑ και θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς και ευγνώμονες γι' αυτό. Τώρα, στην οδηγία για την οποία είμαι εγώ εισηγητής και όπως είπε και ο Σβές, την οδηγία για τις ε, αντισταθμίσεις, για τα συστήματα αντισταθμίσεων για τους επενδυτές και αυτή έχει κολλήσει. Και μετά τη συζήτηση ίσως για την Τραπεζική Ένωση ε, ξεμπλέξουν κάπως τα πράγματα, αλλά στην περίπτωση αυτή χρήσιμο θα ήταν να προωθήσουμε το θέμα της προστασίας των επενδυτών και το θέμα των θεματοφυλάκων και της ευθύνης τους σε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια τότε ήταν αρνητικό που το αποκλείσαμε από τη συζήτηση, σήμερα όμως ίσως θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ήθελε να λάβει το λόγο για το σημείο αυτό. Βεβαίως. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θα λάβουμε υπόψη μερικές παρατηρήσεις ε, των Ευρωβουλευτών. Σίγουρα θα ξαναεξετάσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα των επιλέξιμων φορέων. Είναι ένα ζήτημα που μας προβληματίζει και μας, γιατί είναι ε, λίγοι είναι οι φορείς αυτή τη στιγμή που δρούν ως θεματοφύλακες και δεν είναι ε, εταιρεία με, την, με τον ορισμό της οδηγίας MIFID, ούτε θα έπαιρναν άδεια με βάση την οδηγία MIFID. Τώρα, ποιο μπορεί να είναι, ποιο είναι επιλέξιμο θεματοφύλακα. Φυσικά, βασικό μα στόχο είναι η προστασία των επενδυτών. Αυτός, ε, αυτή είναι και η κεντρική ιδέα τη ρύθμιση. Πάντω, ε, το MIFID θα είναι ένα κατόφλι που θα πρέπει να περάσουν όλοι. Κεφαλαϊκέ απαιτήσει ε, σε ευθυγράμμιση με την οδηγία για τα, για τα κεφαλικά μέσα και τις οργανωτικέ απαιτήσει για την οδηγία για τις αγορέ χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να είναι ένα κατόφλι, ένα ελάχιστο όριο. Αλλιώς δεν θα μπορεί κανείς να δικαιούται να είναι θεματοφύλακας. Πάντως ω προς το χρονοδιάγραμμα. Η πρόταση ΣΕΚΑ 5 δυστυχώς αναβλήθηκε για κάποιο χρόνο. Ελπίζω τελικά να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το AFMD. Πάντως ε, ελπίζω να προχωρήσει η μεταρρυθμίσεις ε, για τους θεματοφύλακες, πριν οποιαδήποτε μεταρρύθμιση για τις οσεκά, γιατί θα πρέπει να γίνει ευθυγράμμιση για τους ε, θεματοφύλακες. Γιατί δεν μπορεί ιδιώτες ε, των ΟΣΕΚΑ να ε, τυχάνουν χαμηλότερης προστασίας από τους επαγγελματίες επενδυτές της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο προτάξαμε ως προτεραιότητα το θέμα των θεματοφυλάκων είναι ότι ε, έχουμε και σε άλλες συζητήσεις, και σε άλλες, άλλες για τις, τα επενδυτικά ιδρύματα γενικώ και ποιο είναι ο ρόλο του στη συζήτηση για τι σκιώδει τραπεζικέ δραστηριότητε. Και εδώ η συζήτηση είναι ευρύτερη από του ΟΣΕΚΑ. Γιατί έχουμε και άλλα επενδυτικά ταμεία που, που προβαίνουν σε δανεισμό κινητών αξιών. Οπότε η συζήτηση είναι πολύ ευρύτερη και οι διαβουλεύσεις μας παρόλο που θα επικεντρώνονται στο ΣΟΣΕΚΑ, δεν ε, θα αποκλείουν ε, ένα ευρύτερο ε, πεδίο εφαρμογή και μια εμβέλεια που θα ξεπερνά το ΣΟΣΕΚΑ. Και γι' αυτό ε, διαχωρίσαμε τη μεταρρύθμιση και τους θεματοφύλακες και τα αποθετήρια από του ΣΟΣΕΚΑ και το ρόλο των επενδυτικών ταμείων στις σκιώδεις τραπεζικές δραστηριότητες. Αυτά προς το παρόν. Εξετάστε προσεκτικά παρακαλώ το θέμα της επιλεξιμότητας των θεματοφυλάκων και να έχετε υπόψη ότι και από άψη κεφαλαίου και από άποψη οργανωτικών εγγύσεων δεν θα πρέπει να είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι από τα στάνταρ της οδηγίας μη για την αγορά των χρηματοπιστωτικών μέσων. Γιατί θα πρέπει ε, να μπορεί κανείς να είναι υπεύθυνο σε περίπτωση απώλειας. Νομίζω ότι είναι απόλυτο απαραίτητο κάτι τέτοιο. Και τέλος ο εισηγητής μας ο κύριος Γκίγκολτ. Σύντομα, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Φαίνεται πως συμφωνούμε αρκετά. Ευχαριστώ και για τις προτάσεις που έγιναν και από την Αιλίν και τον Σαΐντ και και επίσης από την Ανέτε Γιάνσεν. Να ευχαριστήσω επίσης και νομίζω πως είναι η πρώτη φορά όσο καιρό είμαι στην Επιτροπή που κάποιος στην αρχή μιας ομιλίας τόνισε πως ίσως υπάρχει ίσως υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα ή ειδική σχέση με έναν κλάδο για τον οποίο νομοθετούμε. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ανέτ Γένσεν που ξεκίνησε έτσι την ομιλία της. Ε, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στην Επιτροπή μας και είμαι σίγουρος πως ε, αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι εσύ είσαι η μόνη που αντιλήφθηκε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, είναι φυσιολογικό να το προσεγγίσουμε αυτό με έναν τρόπο που θα είναι ότι θα εξετάσουμε όλα τα διαφορετικά χρηματοοικονομικά κέντρα και λογικό να πάμε και στο Λονδίνο και σε άλλες χώρες θα πάμε και θα μιλήσουμε και την άλλη πλευρά. Τα όργανα εκείνα τα οποία προστατεύουν τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και πέρα από αυτό θα ήθελα να πω πως υπάρχει βεβαίως ένα ζήτημα που έχει μεγάλη σημασία. Στον κόσμο των ΟΣΕΚΑ που υποτίθεται ό,τι αφορούσε τους ε, μικροεπενδυτές βλέπουμε πως πηγαίνουμε σε κάποια προϊόντα τα οποία κανονικά θεωρούνται προϊόντα ε, εναλλακτικών επενδύσεων. Και λογικό είναι, μα γιατί να μην τα εναρμονίσουμε όλα αλλά μιλώντας σε επιχειρήσεις και τους καταναλωτές είμαι πολύ επιφυλακτικός γιατί οι ΟΣΕΚΑ έχουν αποδειχθεί τόσο ε, χρήσιμοι γιατί τους ε, θεωρούν οι καταναλωτές αξιόπιστους και άρα αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και θα πρέπει να μας ανησυχεί εάν κάποιοι εκτός Ευρώπης λένε μα κάτω από αυτό το τίτλο μπορείτε να κανονίσετε πάρα πολλά και διάφορα πράγματα και αρχίζουν να συζητάνε τις δικές τους ε, αυστηρότερες προδιαγραφές. Αυτό τελικά μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Οπότε καλό είναι να μην ακολουθήσουμε. Εάν δεν ε, ακολουθήσουμε λοιπόν ε, την προστασία του μικρού επενδυτή και του λιανικού καταναλωτή, θα έχουμε αποτελεσματικότερη προστασία αλλού και άρα ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Νομίζω λοιπόν εδώ πέρα πως ε, και τα συμφέροντα του χρηματοοικονομικού κλάδου συμπλέουν με τα δικά μας και αυτό πρέπει να γίνει στις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Το σχέδιο έκθεσης ε, θα παρουσιαστεί στις 5 Νοεμβρίου, 22 Νοεμβρίου οι τροπολογίες, εξέταση τροπολογιών 17 Δεκεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή 21 Ιανουαρίου του επομένου έτους. Περνάμε στην επόμενη έκθεση, η οποία είναι ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2011. Η κυρία Μαρίζα Ματίας έχει τον λόγο, η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε εδώ στην Επιτροπή σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Πιστεύω ότι με την οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι όλο ένα και πιο παρούσα είτε για τις ε, ε, θεσμικές προσαρμογές είτε στα διάφορα μέσα που έχουν αναπτυχθεί για να απαντηθεί η κρίση που ζούμε κυρίως ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η έκθεση της ε, ΕΚΤ το του 2011 πιστεύω ότι ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τις αλλαγές ε, που είδαμε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απάντηση στην κρίση και αυτό που ε, ξεκαθαρίστηκε και από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΕΚΤ είναι ότι το έτος αυτό είδαμε σοβαρή οικονομική ύφεση όπως ε, παραδείγματος χάρη είδαμε 1,5% ύφεση της Ευρωζώνης και αυτό σημαίνει ότι είχαμε σημαντική προχώρησε και σε σχέση με το 2010 τώρα σε σχέση με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ. Εγώ πιστεύω ότι εμείς θα μπορούσαμε να δούμε δύο πολύ διαφορετικές περιόδους. Το πρώτο εξάμεινο θα έλεγα ότι η δράση της ΕΚΤ ήταν μια δράση παράλογη θα έλεγα εγώ ή τουλάχιστον δυσανάλογη και το δεύτερο εξάμεινο είχαμε μια διαφορετική στάση και μάλιστα προσπάθησαν να τροποποιήσουν ε, τα όσα δεν έκαναν ε, το πρώτο εξάμεινο. Στο πρώτο εξάμεινο η ΕΚΤ ε, αύξησε τα επιτόκια τον Απρίλιο και τον Αύγουστο και η αύξηση αυτή αντικατοπτρίστηκε ε, στους 50 πόντους βάσης και κατόπιν στα τέλη του έτους είδαμε ότι η ΕΚΤ ε, μείωσε και πάλι τα επιτόκια και ακριβώς στο ίδιο ποσοστό. Το τι έγινε λοιπόν στο πρώτο εξάμεινο παρόλο που ήταν βέβαιο ότι ε, το 2012 ε, είχαμε ε, ουσιαστικά διαφορά σε σχέση με το 2011, σε σχέση με το ποσοστό μεγέθυνσης όμως δυσανάλογα αύξησε η τα επιτόκια γιατί είπε ότι έχει να κάνει με τη συγκυρία, με την αύξηση των καυσίμων κυρίως και έτσι λοιπόν αυτή ήταν μια απάντηση δυσανάλογη κατά την άποψή μου. Στο δεύτερο εξάμεινο είδαμε μια απόπειρα αλλαγή τάσης και κυρίως με τη μείωση των επιτοκίων όμως παρόλα αυτά υπάρχει πρόβλημα με την επεκτατική πολιτική της ΕΚΤ στο δεύτερο εξάμεινο και είναι το εξή. Αν ε, δούμε προσεκτικά την ετήσια έκθεση, αυτή η πολιτική δεν είχε αντίκτυπο στην ε, αύξηση ε, των εσόδων ούτε των επιχειρήσεων ούτε των οικογενειών, στην αύξηση της πίστος, της πίστοσης σε αυτούς και λόγω της ε, πολιτικής λιτότητας ε, και της μείωσης των μισθών. Και ακριβώς και γι' αυτό, λόγω της ε, ανεπάρκειας των επεκτατικών πολιτικών, του δεύτερου εξαμήνου, εγώ νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε δύο τεινά σε δύο κυρίες συζητήσεις. Καταρχήν, πρέπει να συζητήσουμε την ίδια την εντολή της ΕΚΤ. Και να δούμε αν είναι λογικό η ε, εντολή της ε, ΕΚΤ ε, να καλύπτει και το θέμα του πληθωρισμού ανεξάρτητα από τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει για την αύξηση των θέσεων Και θα δώσω ένα παράδειγμα για να αντιμετωπίσουμε την τελμάτωση της κρίσης θα έπρεπε να αυξηθούν οι μισθοί στις χώρες της Ευρωζώνης και μάλιστα γιατί με την αύξηση αυτή θα μπορούσαμε να έχουμε ε, την αύξηση της ζήτηση στην Ευρωζώνη και θα μειώνονταν ε, οι ανισορροπίες μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας που βλέπουμε ότι είναι ολοένα και πιο έντονες στα πλαίσια της κρίσης. Αυτό είναι το θέμα της πρώτης της συζήτησης. Η δεύτερη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε έχει να κάνει το τι κάνει η ΕΚΤ πέρα από την εντολή της. Και αυτό σχετίζεται με τις πολιτικές λιτότητας που βιώνουμε σήμερα. Εγώ νομίζω ότι όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής, όπως και εγώ, γνωρίζουν πολύ καλά το ρόλο διαδραμάτισε η ΕΚΤ ε, στην ε, σύσταση μέτρων στα κρατη και για τη δυσιονομική πολιτική και μέτρα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και με συστάσεις ό,τι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες για θέματα ιδιωτικοποιήσεων, φορολογίας κτλ. Υπήρξε λοιπόν μία σειρά συστάσεων που δόθηκαν από την ΕΚΤ στα κράτη-μέλη σε ένα πλαίσιο που εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε δημόσιες πολιτικές πρόθεσης της ανάπτυξης και κάτι τέτοιο δεν προωθήθηκε. Και για να ολοκληρώσω πιστεύω ότι πρέπει να προσεγγίσουμε και ορισμένα άλλα στοιχεία για την ίδια τη λειτουργία της ΕΚΤ. Και εδώ υπάρχουν δύο θέματα που θέλω να τονίσω, δεν θα είμαι εξαντλητική βέβαια. Το πρώτο έχει να κάνει με την απουσία γυναικών στο Δικαιωτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αυτή είναι μια συζήτηση που έλαβε χώρα σε αυτή την Επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το στοιχείο γιατί ε, ουσιαστικά δεν σέβονται καθόλου την ισότητα ε, των ε, δύο φύλων και μάλιστα μέσα στην ίδια την ΕΚΤ. Και δεύτερη, το δεύτερο θέμα είναι η λειτουργία της ΕΚΤ και αυτή έχει να κάνει με το πιο κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει όλο ένα και περισσότερο. Εμείς πρέπει να έχουμε υπόψη τις διάφορες απόπειρες που υπάρξουν για να παραγωνιστεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπου εμπλέκεται η ΕΚΤ. Και εγώ νομίζω ότι έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ ο δημοκρατικός έλεγχος ε, της ΕΚΤ. Υπάρχουν ε, και δύο θέματα που έχουν να κάνουν με τη σημερινή πολιτική και νομίζω ότι επίσης πρέπει να συζητηθούν και να προσεγγιστούν στο πλαίσιο της εκθέσης αυτής. Το πρώτο που θα ήθελα να συζητήσω με τους συναδέλφους είναι αν ε, θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε χωρίς ε, η ΕΚΤ να στέλνει κάποια ε, ξεκάθαρα μηνύματα σε σχέση με την επεκτατική οικονομική πολιτική, νομισματική πολιτική και όχι με κατακραματισμένη πολιτική. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το αν μπορούμε να συνεχίσουμε με μία ΕΚΤ που δεν θα διασφαλίζει σταθερότητα των τιμών. Υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες λοιπόν, ε, όμως αυτή είναι μια πρώτη παρουσίαση ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με την ΕΚΤ και εγώ φυσικά θέλω να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και για αυτά τα ζητήματα αλλά και για άλλα ζητήματα που δεν ανέφερα για να μπορούμε στη συνέχεια να επεκτείνουμε και τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Συγγετρία. Και πάλι έχουμε παρόντες πέντε σκιώδεις ηγητές. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Η κυρία Πέλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτριά μας γιατί μας έκανε μια πολύ τεκμηρωμένη και μεστή παρουσίαση. Και νομίζω ότι το 2011 και από οικονομική και από δημοσιονομική άποψη ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Βέβαια δεν ήταν η πρώτη τέτοια δύσκολη χρονιά, ούτε θα είναι και η τελευταία δυστυχώς. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα ότι αυτό το πρόβλημα θα μας ταλανίσει για αρκετό καιρό ακόμη και θα πρέπει και η λύση που θα προκρίνουμε να έχει αυτή, αυτό το μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πιστεύω ότι και το θέμα της εντολής θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο διεξοδικά. Το 2011 ε, διαιρέθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση είχαμε κάποιες αντιφατικές κινήσεις. Η ΕΚΤ ε, ε δρούσε με έναν τρόπο το πρώτο εξάμεινο, το δεύτερο εξάμεινο με τον αντίθετο. Φαντάζομαι υπήρχαν λόγοι για αυτές τις αντιφάσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και κάποιος προβληματισμός και ανησυχία. 50 ποσοστία της μονάδας είχαμε αύξηση κατά το πρώτο εξάμεινο και ενώ το δεύτερο εξάμεινο είχαμε αντίστοιχη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης. Θα πρέπει λοιπόν να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, να βαθύνουμε στο θέμα και να δούμε πού οφείλονταν αυτές οι αντιφατικές ενέργειες, ποιοι ήταν οι λόγοι για τα βαθύτερα αίτια. Έχαμε και την απόφαση του Δεκεμβρίου και ε, δυστυχώς τα πενιχρά αποτελέσματα από αυτήν. Το 2011 ένα άλλο πρόβλημα που ανέκυψε ήταν το δημοσίου χρέους. Πολύ σημαντικό ζήτημα που επηρέασε και τις τράπεζές μας. Δημιουργήθηκαν προβλήματα και στις τράπεζες και η δημοσιονομική κατάσταση ε, και η χρηματοπιστωτική επιδεινώθηκε. Ήταν αρκετά δραστήρια η έκτα από την άποψη. Υπήρξε το θέμα της αναδιάθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους και είχε πει τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν θα διέγραφε το χρέος. Θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε αυτή την άποψη, ιδιαίτερη από το φως των τελευταίων εξελίξεων και να εξετάσουμε κατά πόσο ήταν καλά τεκμηριωμένη η άποψη της ΕΚΤ τότε. Τον Αύγουστο του 2011 δημιουργήθηκε μια νέα τάση που δεν αφορούσε αποκλειστικά την ΕΚΤ, αλλά είχε περισσότερα σχέση με την εντολή για την ε, πιστοτική πολιτική. Από τον Αύγουστο και μετά ε, υιοθετήθηκε μια πιστοτική πολιτική που είχε αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα για τα πιο περιφερειακά κράτη της Ευρωζώνης και τη δυνατότητα δανειοληψίας τους. Πολλές ήταν οι προκλήσεις, πολλές επικρίσεις επίσης ε, ακούστηκαν εκείνη την εποχή. Στο μεταξύ βέβαια είχαμε μια μετάθεση αυτών των δραστηριοτήτων η δυνατότητα αγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά υπήρξε κάποια μεταστροφή, αλλά καλό θα ήταν να μελετήσουμε όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες και πραγματικά ε, έχω πολλά ερωτηματικά, έχουν μείνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα που χρήζουν διαλεύκασης. Κάτι άλλο που ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εισηγήτρια αφορά το ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΚΤ. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτό το θέμα και να έχουμε μια εκτενή συζήτηση. Ε, αξιολόγηση των κινδύνων, πολιτική για τους κινδύνους, οικονομική ανάπτυξη, ποιε είναι οι προοπτικέ, ποιε είναι οι προκλήσει για την Ευρωζώνη, δυνατότητε διεύρυνση και ούτω καθεξής. Και επίση ε, το θέμα τη εμπιστοσύνη προ την ΕΚΤ και την, ε, το θέμα του δίκτυου εμπιστοσύνη. Τέλος, ε, σημαντικό όμως θέμα, τι συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες. την τελευταία ολομέλεια είχαμε σχετική συζήτηση. Εποπτικές αρμοδιότητες της ΕΚΤ και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τους, κατά πόσο θα σκόπιμο κάτι τέτοιο και τα συναφή ζητήματα. Είχαμε και την ε, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την, ε, της έκθεση του 2010 της ΕΚΤ συγκρίνοντας τις δύο εκθέσεις βλέπουμε ότι έγινε μία μεταστροφή στις προτεραιότητες. Το 2010 είχαμε κάτι, κάποια σημεία, κάποια θέματα που θεωρώνται σημαντικά που παραλείπονται πλήρως από την έκθεση του 2011. Στο σημείο 13 για παράδειγμα αναφερόταν η πρόταση της θέσπισης ε, της ε, δημιουργίας ενός ιδρύματος ε, για την αξιολόγηση των πιστώσεων. Τελικά αυτό κατέπεσε αυτή η, η πρόταση. Ίσως σκόπιμο θα ήταν να τη μελετήσει η συγγήτρια και να δει γιατί να βάγισε. Κρίθηκε ασήμαντη ή αναποτελεσματική. Ας το κοιτάξουμε και αυτό. Πάντως προσβλέπω σε στενή συνεργασία με την εισηγήτρια. Την ευχαριστώ για το μέχρι τώρα έργο της και ελπίζω να λάβετε υπόψη και τις τροπολογίες που θα καταθέσω. Ο κύριος Χουάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος που για το θέμα αυτό ε, θα συνεργαστώ με γυναίκες που είναι οι σκιώδεις συγγήτρες και οι συγκήτρια και να ευχαριστήσω θερμά την ε, Μαρίζα. Πήγαμε μαζί στην Φραγκφούρτη, στην πρώτη μα επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είχαμε πολύ σοβαρέ συζητήσει με εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Τράπεζας. Ε, το θέμα τη περιορισμένη επαναγορά ε, ομολόγων, τριετών ομολόγων που είχε αναγγείλει η ΕΚΤ αγορά ομολόγων ε, για χώρες που θα ενταχθούν στον μηχανισμό σταθερότητας και μιλήσαμε και για την κεντρική εντολή ε, που διαπιστώσαμε ότι μερικές φορές ε, ξεπερνούσε την απλή εντολή της σταθερότητας των τιμών γιατί ε, ασχολήθηκε και με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και με δημοσιονομική πολιτική, κάτι που αρχικά δεν ανέπιπτε στην εντολή της και στον τομέα αρμοδιοτήτων της. Η έκθεση αυτή εξετάζεται σε μια πολύ ιδιάζουσα στιγμή, γιατί ξέρετε ότι σήμερα έχει ανακύψει και το πρόβλημα του δημοκρατικού ελέγχου της δημοσιονομικής διακυβέρνησης αλλά και της νομισματικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και όχι μόνο της Ευρωζώνης γιατί η συζήτηση αυτή ε, θα επεκταθεί και στο θέμα της ε, δημιουργίας, της μελλοντικής δημιουργίας της Τραπεζικής Ένωσης. Οπότε, επ' ευκαιρία αυτής της έκθεσης θα υποβάλουμε διάφορα ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα LTRO. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κινητό κοντά σας ενεργοποιημένο γιατί υπάρχουν παρεμβολές στο μικρόφωνο ή να αλλάξετε θέση. Sorry everybody, but it's a good idea if we can hear. Λυπάμαι, αλλά καλύτερα να ακούγεται ο μιλητής. Για το πρόγραμμα LTRO. Ε, πάνω από 500 τράπεζες συμμετείχαν στο πρώτο πρόγραμμα έκδοσης, με βάση το οποίο η ΕΚΤ μέσα τρία χρόνια, με 1% ε, επιτόκιο για τρία χρόνια, δάνεισε περίπου 500 δις. Ε, και μάλιστα ε, θα εξεταζόταν η πρόταση αυτή και αργότερα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή η ρευστότητα από τις τράπεζες για να μειωθεί η πίεση προς τα κράτη και ένα τμήμα της ρευστότητας τελικά τοποθετήθηκε στις ε, τράπεζες από την Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια θα πρέπει να διαρωτηθούμε, ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο. Βέβαια έγινε ε, μια διατησία από την Κεντρική Τράπεζα μεταξύ του LTRO και του SMP του προγράμματος δηλαδή εξαγοράς δημοσίου χρέους ε, των χωρών που υπέστησαν κερδοσκοπικές ενέργειες. Επίσης, το... Ε, επίσης, αναφέρθηκε το θέμα της κερδοσκοπίας. Πώς θα την εντοπίσουμε, πώς θα πρέπει να δώσουμε άδεια τραπεζικών δραστηριοτήτων στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας από τη στιγμή που θα έχουμε τον έλεγχο των πιστώσεων που δόθηκαν, των δανείων που δόθηκαν για να βοηθήσουμε τις χώρες ε, που υπέστησαν την κερδοσκοπία. Βέβαια, υπήρχε ένα πρόβλημα ως προς την ε, ιδέα αυτού του θέματος και ε, διαρωτόμαστε ποια είναι η θέση της ΕΚΤ ε, ως πιστωτή. Η, όσον αφορά την Ελλάδα, από τις αρχές του 2010 η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικά ομόλογα ε, περίπου 500 δις ονομαστικής αξίας. Βέβαια, με τη διακύμαση των ομολόγων και της απώλειας της ονομαστικής του αξίας, τελικά η ΕΚΤ πλήρωσε πάνω, λιγότερο από 40 δισεκατομμύρια για να τις αγοράσει. Βέβαια, ε, αρχίζουν να γίνονται λεξιπρόθεσμα αυτά τα ομόλογα και η εκδικεί την ε, τιμή που πλήρωσε. Άρα έχει μια υπεραξία γύρω στα 11 δισεκατομμύρια εις βάρος της Ελλάδας χωρίς να συνυπολογίσουμε και τους στόκους. 11 δισεκατομμύρια είναι πάνω από, τα, 4% του ελληνικού ΑΕΠ. Δηλαδή τέτοιου ίδιες υπεραξίες θα πραγματοποιούσε η ΕΚΤ με βάση τις ε, συνθήκες της αγοράς. Δεν νομίζω. Και μάλιστα τελικά την ενθάρρυνε αυτή την κατάσταση η ΕΚΤ, γιατί απέκλεισε από την, αποκλείστηκε η ΕΚΤ από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους στις αρχές του 2012. Ενώ 96% ε, των ε, πιστωτών, των ιδιωτών πιστωτών αναγκάστηκαν ε, να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, ενώ η ΕΚΤ αυτό αποκλείστηκε από αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, 3,6 δισεκατομμύρια είχε αύξηση ε, ως προς στην ίσπραξη των τόκων, εξηγώντας ότι οι διαφορές αυτές σε σχέση με το 2010 προερχόταν από το πλαίσιο του S&P. Οπότε καταλήγουμε σε ένα παράδοξο. Ένα μεγάλο τμήμα των ενισχύσεων προς την Ελλάδα ουσιαστικά βοήθησαν να ε, βελτιώσουν τον ισολογισμό της ΕΚΤ χωρίς ε, ούτε η ελληνική οικονομία, ούτε η πραγματική οικονομία, ούτε η Ελλάδα να δρέψει τους καρπούς αυτής της βοήθειας και χωρίς καν να, αγγίξει, να αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο παράδοξο, οπότε πολλά ερωτηματικά υπάρχουν για τη δράση της ΕΚΤ, ειδικά για την πλούσια σε γεγονότα χρονιά το 2011. Γι' αυτό και προσβλέπω σε πολύ καρποφόρα συζήτηση με την εισηγήτρια και τους λοιπούς και όδης εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σάρον. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, επομένω δεν θα μακρηγορήσω. Καταρχήν ήμουν εισηγητή ε, για την έκθεση τη ε, ΕΚΤ ε, πέρσι, έτσι λοιπόν χρειάζεσαι Μαρίσα βοήθεια. Ευχαρίστω να είμαι σε αυτή την ισορροπημένη ομάδα από άποψη συμμετοχή των δύο φίλων και να συζητήσουμε αυτή την έκθεση ΕΚΤ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Μπέρναρ Λάγκεν πριν ένα έτος σε αυτό τον οίκο όταν ε, πέρσι το καλοκαίρι έφυγε, άρχισε να αγοράζει τα ισπανικά και τα ιταλικά ομόλογα, είπε. Φυσικά, χωρίς την παρέμβαση της ΕΚΤ θα ήταν χειρότερη κατάσταση. Και αυτή την εντύπωση έχω, χωρίς ε, τις παρεμβάσεις, ε, τις περσινές της ΕΚΤ και των τελευταίων μηνών θα ήταν χειρότερη η κατάσταση. Και τώρα, εγώ ως Ευρωπαίος υπέρ της Ομοσπονδίας μου λείπει καθημερινά ένας ε, ε, υπουργός οικονομικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ένας ταμείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να κάνουν ε, όλο αυτό το έργο που αναγκάζεται να κάνει η ΕΚΤ τώρα. Έτσι λοιπόν αυτή η συζήτηση για το ρόλο της έκθεσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και για την αποτελεσματικότητα ε, των μικροπρόθεσμων αναχρηματοδοτήσεων. Είναι καλή σύμπτωση που η πρώτη μικροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση έγινε πριν ε, ε, τα Χριστούγεννα ήταν τα κάλαντα της έκτη για τα τελευταία Χριστούγεννα. Άρχισε να αγοράζει ομόλογα και να δίνει χρήματα σε ισπανικές τράπεζες για να αγοράσουν ισπανικό χρέο. Όμως τώρα ήρθε ο καιρό να αναλύσουμε το αποτέλεσμα ε, αυτών των ε, συναλλαγών γιατί μετά από το δεύτερο ελτιρεού το Μάρτιο φέτος είδαμε ότι δεν ρεεί η πίστοση από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Και επίση ο κ. Δράγκη αναγνώρισε εδώ στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή ότι τώρα η αποτελεσματικότητα των αναχρηματοδοτήσεων δεν είναι καλή και μπορούμε στην Ισπανία να μιλήσουμε για ένα αποτέλεσμα ε, συγκέντρωσης, δηλαδή θα αγοραστεί δημόσιο χρέος, θα τα κονδύλια χρησιμοποιηθούν όλα για να, για να αγοραστεί δημόσιο χρέος και δεν θα ε, διοχετευτούν ε, στα νοικοκυριά ή στις επιχειρήσεις. Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι το εξή. Εγώ πιστεύω στο ευρώ. Το 2010 όταν ε, συζητήσαμε τη δέση μέτρων για την ε, χρηματοοικονομική υποπτία, εγώ ήθελα να πω στο ευρώ που εμπιστεύομαι και στην έκτη που εμπιστεύομαι στο τέλος ε, της ομιλίας μου και είμαι υπέρ ενός ανεξάρτητου νομίσματος, κοινού νομίσματος, έτσι λοιπόν θα επικεντρώσω τη συζήτηση στο σε ένα διπλό σύστημα. Χαίρομαι που στη φετινή έκθεση υπάρχει ένα κεφάλαιο της ΕΚΤ ε, που ε, έχει να κάνει με το σύστημα με τους δύο στόχους ε, και φυσικά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό για τις συζητήσεις που θα έχουμε σε αυτό τον νοικό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο στην περσίνη έκθεση και έπρεπε να δούμε ε, αυτές τις ε, ροές να είναι σε κάποια άλλα έγγραφα και όχι στην έκθεση της ΕΚΤ. Εγώ θα ήθελα να έχουμε μια βιώσιμη νομισματική ένωση και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια που από κάποιες εθνικές κεντρικές τράπεζες πηγαίνουν σε άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες και αναρωτιέμαι αν αυτές οι ενισορροπίες είναι βιώσιμες και να γίνονται μόνιμες ή όχι και θα πρέπει να αναλύσουμε πώς ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, η Federal Reserve και η δική τους κεντρική τράπεζα ασχολείται με τα ζητήματα αυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό. Και επίσης ε, ενδιαφέρομαι να μελετήσω την κατάσταση ορισμένων εθνικών κεντρικών τραπεζών όπως έκανε η Ισπανία για την ε, έκτακτης ανάγκης βοήθεια ρευστότητας θα είναι ευκαιρία να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Και επίση χαιρόμαι που ο κύριο Δράγκη είναι τώρα πρόεδρο τη ΕΚΤ, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ ικανό άνθρωπο με εμπειρογνωμοσύνη και πολλέ γνώσει και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση προ το συμφέρον των πολιτών μα και του μέλλοντό μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Σβέν δεν είναι εδώ. Φιλίπ, φαντάζομαι τον αντικαθιστά. Ούτε ο Σβέν, ούτε η Εύα ότι η Εύα υποτίθεται πως θα ήταν εδώ. Θα πω λοιπόν ένα πράγμα για να μην επαναλάβω όλα όσα ακούστηκαν. Σύμφωνο πολλά από αυτά, αλλά για το γεγονός πως η ΕΚΤ ε, φαίνεται πως είναι έτοιμη να αναλάβει και άλλες ε, εξουσίες πέρα από τις ήδη πάρα πολλές που έχει, θα έλεγα πως θα πρέπει να ξαναδούμε το πώς γίνονται αυτές οι εκθέσεις και το αν θέμε να τις αναβαθμίσουμε. Γιατί το ζήτημα της δημοκρατικής νομοποίησης των όσων κάνει η ΕΚΤ είναι πλέον σοβαρό και αν κάνουμε μια έκθεση σήμερα ίσως από του χρόνου θα πρέπει να κάνουμε δύο εκθέσεις όταν η ΕΚΤ θα είναι και εποπτική αρχή και πρέπει να κάνουμε δύο χωριστές θεωρώ εγώ για να έχει και διαφορετική στάση η ΕΚΤ όταν έρχεται για τη μία έκθεση και όταν έρχεται για την άλλη. Και δεν θέμε να τα μπερδεύουμε. Αλλά ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα στην ΕΚΤ πως πράγματι αναμένουμε από αυτούς και όχι απλά τους ζητάμε να είναι υπόλογοι θεωρούμε πως ε, αυτό πρέπει να ε, κάνουμε και από τώρα ήδη εν είδη προειδοποίησης. Πρόεδρος, ε, να απαντήσω και σε αυτό, να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι πρέπει να κάνουμε την ετήσια έκθεση, όπως κάνουμε για τον ανταγωνισμό, από τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Και βεβαίως και λόγω του ρόλου μας στη λογοδοσία της ΕΚΤ, Νομίζω πως είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό με τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Ειδικά αν ε, χρειαζόμαστε περισσότερη λογοδοσία όσον αφορά τις προτάσεις ε, Τραπεζικής Ένωσης και ελπίζω οι συνάδελφοι να ενημερώσουν τους πρόεδρους των ομάδων τους έτσι ώστε όταν την επόμενη φορά ξαναζητήσουμε να ληφθεί υπόψη αυτό το ζήτημα ίσως οι πρόεδροι ομάδων συνειδητοποιήσουν πως η δημοκρατική λογοδοσία το απαιτεί. Ο Ντέρκ, κατόπιν ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην έκθεση, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο το 2010 επένεσε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τα όσα έκανε κατά τη διάρκεια της κρίσης και δεν έχουμε πολύ, όπως και φέτος ε, θα θεωρήσει το Κοινοβούλιο πώ έκανε εξαιρετική δουλειά η Κεντρική Τράπεζα. Έχω να κάνω όμως τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η ε, πράξη μαξοπρόθεσμη χρηματοδότησης του 2011 και 2012 έδωσε γύρω στο 1-3 εκατομμύριο ευρώ φτηνών πιστώσεων σε πιεζόμενε τράπεζες στα κράτη-μέλη. Όμως δεν επέτυχε τον σημαντικότερο στόχο του, δηλαδή να αυξηθεί ο δανεισμό σε επιχειρήσει και νοικοκυριά. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντί για τρία χρόνια επέτυχε μόνο τρεις μήνες σταθερότητας της αγοράς. Επίσης αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο μπαζούκα της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή είναι διατεθειμένη να αγοράσει απεριόριστο δημόσιο χρέος βραχυπρόθεσμο βεβαίως. Ε, η απόφαση αυτή ενέχει κινδύνους. Να υπενθυμίσω πως η Γερμανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα καταψήφισε αυτή την απόφαση και την προηγούμενη εβδομάδα. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο θεώρησε πως μια τέτοια πράξη θα ήταν ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο. Και εγώ συμφωνώ και με την ε, Γερμανική Κεντρική Τράπεζα και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Βεβαίω υπάρχει και ο κίνδυνος του ηθικού κινδύνου. Προσφέρεται να αγοράσει απεριόριστα ομόλογα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα υπό τον όρο πώς θα συμφωνήσουν με το χρονοδιάγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής οι χώρες. Αλλά πώς θα μπορέσει να το επιβάλλει αυτό. Θα τραβήξει το χαλί κατά από τα πόδια τους εάν δεν συμμορφωθούν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί μόνο να ελπίζει πως οι απρόβλεπτες πολιτικές αποφάσεις στα κράτη-μέλη θα κυλήσουν όπως θέλει εκείνη. Ο κίνδυνος είναι πως οι χώρες θα χαλαρώσουν, όπως έχει ήδη συμβεί, και δεν θα έχουν κίνητρο για γρήγορες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα καταστεί έτσι ακόμη πιο μακροπρόθεσμη η κρίση. Και δεύτερον, ο ισολογισμός της ήδη είναι προβληματικός, ένα τρίτο του είναι στην περιφέρεια και το ερώτημα είναι αν η Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα μιας χώρας η οποία δεν μεταρρυθμίζει. Αν δεν το κάνει θα πανικοβληθούν οι αγορές. Τι σκοπεύει ακριβώς λοιπόν να προλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα συσσωρεύσει χρέος το οποίο δεν θα πληρωθεί και θα γίνει η ίδια μία α, τράπεζα η οποία δεν θα είναι βιώσιμη και δεν είναι πλέον ο δανειστής τελευταίας καταβηγής, αλλά αντιθέτως είναι ο δανειστής ο οποίο στρέφονται πρώτα όλοι και τώρα παίζει πολιτικό ρόλο με το να επιτηρεί τη χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους. Μα η κεντρική τράπεζα δεν είναι κεντρική κυβέρνηση. Μπορεί να τυπώσει χρήμα, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει δουλειέ. Δεν μπορεί να προωθήσει μεταρρυθμίσεις. Αυτό πρέπει να το κάνουν οι πολιτικοί. Αλλά αυτοί φοβούνται τους ψηφοφόρους τους. Και τέταρτον και τελευταίον υπάρχει και το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Στο ευρωσύστημα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θεσμικό όργανο το οποίο λειτουργεί σαν το Βατικανό. Δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Τα πρακτικά των κονκλαβίων είναι μυστικά. Και δεν υπάρχουν και γυναίκες από πάνω. Ε, είδατε που συμφωνούμε σε κάτι. Ο δε πρόεδρος της, ο κύριος ε, Ντράγκη, είναι πλέον Πάπας συναντάει τους διάφορους καρδιναλίους στην Φραγκφούρτη, η οποία έχει γίνει η νέα Ρώμη της Ευρωζώνης. Οπότε, όταν βρίσκεται στο μάτι του πολιτικού κυκλώνα και όταν θα βρεθεί στο μάτι του πολιτικού κυκλώνα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ανθρώπους οι οποίοι δεν την γνωρίζουν και θα είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο δεν θα έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Και νομίζω αυτός είναι ένας τεράστιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή γιατί η ΕΚΤ έχει γίνει ο ε, κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας. Ναι, όντω. Μια και οι πάπε, <laughs> αν οι πάπε είναι μόνο άντρε, αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Η Σιλβή. Εγώ δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να ε, πατήσω ένα αστείο. Ξέρετε γιατί, όπω είδαμε μερικοί, Ευρώπη έχει προβλήματα γιατί ε, ένα Γερμανό βρίσκεται επικεφαλή του Βατικανού και ένα ε, Ιταλό επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι ο λόγο. Εν πάση περιπτώσει. Ε, Όντω, ε, η, η δράση τη ΕΚΤ ήταν σε μια δύσκολη περίοδο αξιέπαινη. Καταρχήν, είχαμε τα γεγονότα. Αν σκεφτούμε τι συνέβη το 2011, συνειδητοποιούμε ότι μερικές αποφάσεις ε, ε, χρειάστηκε να ληφθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε με το περιεχόμενο. Αναφέρθηκαν από το ΛΙΑΜ, κρίση του ευρώ και το καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν με την απόσταση που μας χωρίζει πια και με ψυχραιμία να κάνουμε μια αποτίμηση της κατάστασης και να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Ε, επίσης, το 2011, όπως είπαν μερικοί, στα τέλη του 2011, η Κούντρουν Τουρούμπερ Γούγκερελ, που ήταν η μοναδική γυναίκα ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρετήθηκε και η μάχη που δίνουμε τώρα για να εξασφαλίσουμε μια ελάχιστη ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, ε, προσπαθεί να διορθώσει μια κατάσταση που δημιουργήθηκε εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου ξεκίνησε μια καινοτόμα πρωτοβουλία, αξιέπαινη, γιατί πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης έχουμε μια απόπειρα για μια σφαιρική προσέγγιση. Και αντί να επιλέγουμε μεμονωμένες ε, λύσεις ε, και κατακαιρματισμένες, τελικά η ε, αρχή κρατών και κυβερνήσεων ασχολήθηκαν όχι μόνο με το δημοσιονομικό θέμα, αλλά και με το τραπεζικό, το οικονομικό, της δημοκρατίας και της λογοδοσίας, accountability που δεν υπάρχει μετάφραση στα γαλλικά, ενδιαφέρον και αυτό. Τώρα, το θέμα είναι πώς μπορούμε ε, να έχουμε αυτή την εργασία εξακρίβωσης του τι συνέβη και ελέγχου. Νομίζω ότι από εμά εξαρτάται να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Ραμόν αλλά και οι του ΕΛΚ θα φροντίσουν γι' αυτό. Ανάγκη ε, να εξακριβώσουμε πώς ανταποκρίνεται η ΕΚΤ ε, στις ε, αρμοδιότητές της. Και αυτό είναι ο μύτος Αριάδης, να δούμε ποιες είναι οι δραστηριότητες της ΕΚΤ και νομίζω ότι η συγγήτρια θα το λάβει αυτό υπόψη. Άλλωστε η έκθεση αυτή δεν είναι η ευκαιρία για να τροποποιήσουμε την εντολή της ΕΚΤ. Εμείς υποχρεώμαστε να εφαρμόσουμε τις συνθήκες και να συμμορφωθούμε με αυτές. Έτσι μόνο θα ενισχύσουμε την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων. Μπορεί για το μέλλον να εκφέρουμε μια επιθυμία για κάποιες αλλαγές, γιατί θα έχουμε και την έκθεση της Μαρία Τίσεν που θα λάβει υπόψη κάποιες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το μέλλον, αλλά να αποφύγουμε πληθώρα σχολείων και κριτικών που μπορεί να ικανοποιούν τους μένει τους δε, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε μια έκθεση για την ανάλυση και τη, της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι τελευταίες προτάσεις είναι καινοτόμε και οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ε, θα στενιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τραπεζική Ένωση είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι αυτή η ετήσια έκθεση το, η σωστή ευκαιρία και η κατάλληλη ευκαιρία για να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ και επανέρχομαι στην εισηγήτριά μας. Οι διερμηνείς θα μας δώσουν ένα δεκάλεπτο ακόμη, γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο και θέλουμε να προλάβουμε να εξετάσουμε και την έκθεση του Γκένερ Χόκμαρκ. Παρακαλώ λοιπόν ε, προσπαθήστε να είστε σύντομοι, παρόλο που είναι πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τα σχόλια που έκαναν οι προσωπώντες ομάδες τους. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και δεν διαπίστωσα σημαντικές διαφωνίες σε ό,τι αφορά τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσής μου. Δεν πρόλαβα να ασχοληθώ με όλα τα ζητήματα που θα πραγματεύομαι στην έκθεσή μου. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε κάποια θέματα που θα πρέπει να εμβαθύνουμε Ξεκινώ από την τελευταία παρέμβαση, το θέμα της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, πέραν της ανάγκης να είμαστε ε, αυστηροί ε, και να εμείνουμε στην εντολή μας, ε, δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη. Το 2011 η ίδια η ΕΚΤ επανειλημμένως παρενέβη την εντολή της. Το είπε και ε, ο πρώτος και ο που μίλησε για το θέμα αυτό. Αναγκαστικά υπάρχει μια αλληλεπίδραση των δύο θεμάτων. Γιατί όντως ε, οι συνθήκες ε, περιχαρακώνουν την εντολή της ΕΚΤ και εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε τις συνθήκες, αλλά η ΕΚΤ μερικές φορές ξεπερνά την εντολή της. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε για την ανάγκη να ενισχυθούν ε, τα μέσα δημοκρατικού ελέγχου και να δούμε πώς ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβάλει προτάσεις που θα λαμβάνονται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το θέμα της δημοκρατικής νομοποίησης, της αποτελεσματικότητας ή όχι των μακροπρόθεσμων αναχρηματοδοτήσεων, το θέμα της ε, νομοποίησης ε, κατά πόσο είναι θεμητή η υπεραξία που δημιουργεί η ΕΚΤ αγοράζοντας ε, ομόλογα ε, χωρών που βρέθηκαν στον διχονισμό της διάσωσης και τα τεράστια κονδύλια που έδωσε αλλά και που κέρδισε. Όλα αυτά τα θέματα θα τα λάβω υπόψη στην έκθεση. Θα σας στείλω στο τέλος της εβδομάδας το προσχέδιο και μην ξεχνάτε ποια είναι η τελική προθεσμία για τις τροπολογίες για να τις καταθέσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το σχέδιο έκθεσης ε, έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου, τροπολογίες 25 Οκτωβρίου, συζήτηση επιτροπολογιών 19 Οκτωβρίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 21 Ιανουαρίου και ελπίζουμε ότι θα πάει στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Έτσι λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στην έκθεση του κυρίου Χόκμαρκ. Έχουμε την πρώτη συζήτηση για τα επιστοτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ναι, και το πλαίσιο για την ε, εξυγίανση και την αναδιάρθρωση την ανάρθρωση. Λυπάμαι που δεν έμεινε πολύ χρόνο. Ε, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να σου δώσουμε και περισσότερο χρόνο στο μέλλον. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ. καθώς ε, έχουμε περιορισμένο χρόνο για την έκθεση αυτή και λυπάμαι. Νομίζω ότι είναι όρθο να πούμε ότι ζούμε δύσκολους καιρούς και αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις. Ε, ε, δύσκολο γιατί όλοι βλέπουμε τις συνέπειες όταν οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στο πλήρη δυναμικό τους. Υπάρχει αντίκτυπο στην οικονομία, αλλά έχουμε και προκλήσεις γιατί πρέπει να λάβουμε όχι μόνο αποφάσεις, αλλά πρέπει να λάβουμε και τις σωστές αποφάσεις ε, που σε μακροπρόθεσμη προοπτική να μπορούν να καταστήσουν ισχυρή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, έχω ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας. Και νομίζω ότι πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίω όχι η Κίνα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Αλλά δεν έχουμε τη μεγαλύτερη αγορά. Και από τη δική μου σκοπιά, είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις να διασφαλίσουμε αυτή, δηλαδή ότι θα κρατήσουμε ενωμένη την Ένωση, να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό και να αναπτύξουμε τις καλύτερες από τις ε, ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό και την ισχύ της στην οικονομία. Και αυτό ισχύει και στις ευρωπαϊκές ε, χρηματαγορές όπως και σε άλλα σε άλλους τομείς της Ένωσης και νομίζω ότι αυτή είναι η δική μας ευθύνη να το πράξουμε. Νομίζω ότι τα κυρία μέσα για το σκοπό αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα νέο εγχειρίδιο κανόνων που θα καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει να το καταρτήσουμε αυτό το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε την νομοθεσία σχετικά με τις εποπτικές αρχές συζητούμε την έκθεση του κ. Σάιμον ε, σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων και δεν είναι εύκολο αυτό. Ε, το καθήκον μας ε, έχει απασχολήσει καιρό και δεν νομίζω ότι είναι λάθος να πει κανεί ότι μάλλον θα χρειαστούμε και ακόμη περισσότερο χρόνο για να τα ρυθμίσουμε τα ζητήματα αυτά, αλλά το χρειαζόμαστε και έχουμε και τη διαδικασία της μεταρρύθμισης των κεφαλαϊκών απαιτήσεων. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Και τώρα έχουμε τη διαχείριση της τραπεζικής κρίσης ε, με την ανόρθωση και την εξυγίανση. Γιατί και αυτό πρέπει να γίνει, γιατί έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών τραπεζικών αγορών και χρηματαγορών. Και όταν συζήτησα με τους συζητητές, διαπίστωσα ότι όλοι έχουμε προθυμία να πετύχουμε αποτελέσματα. Και είναι ρεαλιστική και αποφασιστική αυτή η επιθυμία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε ενωμένη την Ένωση. Και είναι ισχυρή η πεποίθησή μου ότι θα είναι δυνατό να προχωρήσουμε προς τα μπρος και να ψηφίσουμε αυτή την νομοθεσία. Είναι κάτι θεμελιώδε. Ξέρω ότι έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις, ανεξελίξη για την Τραπεζική Ένωση παράλληλα και είναι εύκολο να πούμε ότι χρειαζόμαστε καλύτερη εποπτεία. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Και έχουμε και πολλά άλλα ζητήματα Όμω, Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν μπορεί κάποιος να φτιάξει τη στέγη χωρίς να έχει τα θεμέλια. Και αν αποτύχουμε, για το σύστημα κατάθεσης εγγύσεων των κεφαλαϊκών απαιτήσεων και την εξυγίανση, την όρθωση και την των τραπεζών, τότε θα έχουμε αποδυναμώσει την Ένωση και θα έχουμε μειώσει τι ευκαιρίες που έχουμε. Έχουμε ευθύνη εδώ για να πετύχουμε αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση της Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην νομοθεσία μας ε, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τις ε, χρηματαγορές και είναι ένας ε, τρόπος να αναζωογονήσουμε τον καπιταλισμό έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί από όλους και από την αριστερά και από το κέντρο και από τη δεξιά. Γιατί το πλήρε νόημα του σημαντικού αντικτύπου αυτή τη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την αδόρφωση και την εξυγίανση είναι ότι οι μέτοχοι θα έχουν την πλήρη ευθύνη Δηλαδή ότι θα πετύχουμε να έχουμε μέσα τα οποία θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι και σημερινές τράπεζες ε, που αποκαλούνται πολύ μεγάλες για να αποτύχουν, μπορούν να αποτύχουν χωρίς ε, να ζημιώνουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα ως τέτοιο. Οι τράπεζες που δεν λειτουργούν σωστά θα πρέπει να μπορούν να εξαφανιστούν από την αγορά. χωρίς να υπάρχει ζημία του χρηματοοικονομικού συστήματος. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να σώσουμε ό,τι είναι δυνατό να σωθεί, αλλά να υποστηρίξουμε και το σύστημα που χρειάζεται οικονομία για να λειτουργήσει. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική στις μελλοντικέ συζητήσεις. Θα ήθελα να διασφαλίσω ότι κάνουμε μία διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών φαινομένων. Το πρώτο είναι όταν έχουμε μία τράπεζα σε κρίση και το άλλο όταν ε, έχουμε μία τραπεζική κρίση. Δηλαδή, αν γενικεύσω, αυτά είναι δύο διαφορετικά προβλήματα. Όταν έχουμε μία τράπεζα σε κρίση, Κυρίως αυτό αποτελεί αποτέλεσμα κακού επιχειρηματικού μοντέλου, κακής ηγεσία, ε, κακή ανάληψη κινδύνων κτλ. Κακής διαχείρισης, κακής διοίκησης και συνήθως χάνονται οι επενδύσεις και οι τίτλοι. Ενώ όταν έχουμε μια συστημική κρίση, μια τραπεζική κρίση, τα προβλήματα έρχονται εξωτερικά, από έξω στις τράπεζες. Κάποιες τράπεζες είναι πιο καλά προετοιμασμένες, ενώ κάποιες άλλες όχι και τόσο καλά. Όμως ε, και πάλι το σοκ ε, ζημιώνει όλο το σύστημα. Λύτει όλο το σύστημα. Και αυτό σημαίνει ότι διαφέρει κάπως η κατάσταση. Οι απώλειες συνήθως είναι δυνατόν να εκπληθούν όταν έχουμε μια συστημική κρίση. Και σε μια συστημική κρίση Νομίζω ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα πράγμα, το φόβο. Ο πρόεδρος Ρουσβελτ κάποτε είπε ότι το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο φόβος. Και ο φόβος είναι το κύριο πρόβλημα σε μια συστημική τραπεζική κρίση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι τα εργαλεία που προτείνει η Κομισιόν είναι σημαντικά δηλαδή ο διαχωρισμός των κακών από τα καλά περιουσιακά στοιχεία, πώληση τραπεζών, ενδιάμεσο ίδρυμα και διάσωση με διαμέσα. Όμως ε, εξαρτάται από τι είδους κρίση μιλάμε και σε ποια κλίμακα βρισκόμαστε. Δηλαδή μιλάμε για μια τράπεζα σε κρίση ή για μια πλήρη κρίση τραπεζών. Επίσης, ε, έχουμε και προσωρινή δημόσια δημόσιες εγγύσεις και σε μια στιγμική κρίση νομίζω ότι είναι πιο αποδεκτό να πούμε κάτι τέτοιο γιατί πιθανότατα όταν ανακάψει η οικονομία θα ανακτηθούν και οι αξίες ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο όταν έχουμε μια και μόνη τράπεζα σε κρίση. Και γι' αυτό είναι από τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω στην Επιτροπή μαζί με του Σκιώδης είναι πώ θα διασφαλίσουμε ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να καταπολεμήσουμε το φόβο. Όταν ε, κανένας άλλος δεν μπορεί να καταπολεμήσει το φόβο στο τραπεζικό σύστημα, τότε το κράτος και οι κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να ευσέλθουν. Και πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στις ε, πιο βαθιές κρίσεις που έχουμε δει στον τραπεζικό τομέα αυτά τα εργαλεία ήταν ζωτικά για την αποκατάσταση της τάξης. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι δεν είμαι και τόσο σοσιαλιστής. Έτσι λοιπόν, όταν μιλώ για προσωρινή δημοσία ιδιοκτησία, δεν είναι ότι βλέπω εδώ ότι είναι των τραπεζών και ένα τέτοιο κύμα. Μπορώ να πω ε, στο, ε, συνάδελφο ε, ότι το αυτό προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ιδιωτικοποίηση μετά την κρίση, όμω πρέπει να υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Πρέπει να καθορίσουμε κάποια σχέδια ε, ανόρθωσης ε, και πρέπει να δούμε πότε θα επισέρχονται οι αρχές. Θα υπάρχει μια έγκαιρη παρέμβαση. Πρέπει να συστήσουμε έναν ειδικό διευθυντή για να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτό θα ήθελα να το συζητήσω με τους ε, σκιώδεις, γιατί μπορεί, παραδείγματος χάρη, η ειδική διοίκηση, ένας ειδικός διευθυντής να είναι και περισσότερο στο τμήμα της εξυγένσης παρά στο θέμα της ανόρθωσης. Θα το δούμε αυτό, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διάσωση με ίδια μέσα, το bail-in λειτουργεί. Είναι σημαντική πρόταση αυτή, αλλά θα ήθελα να πω ότι το bail-in είναι ένα πολύ καλύτερο εργαλείο να έχει κανείς μέχρι να το χρησιμοποιήσει, γιατί όταν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσει, Υπάρχουν άλλα προβλήματα που θα προκύψουν, ε, προβλήματα ε, μετάδοσης μέσω άλλων τραπεζών και άλλων ιδρυμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ε, χρειαζόμαστε να προσθέσουμε και άλλα εργαλεία, αλλά να διασφαλίσουμε ότι το μέσο του Μπέιλιν θα μπορέσει να λειτουργεί και όταν έχουμε μια βαθιά τραπεζική κρίση. Και ξέρω τις συζητήσεις ε, και τις προτάσεις των σκιωδών σε σχέση με το μέσο αυτό του bail-in, δηλαδή διάσωσιμη μέσα και είπαμε την επικοδομητικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε τι θα κάνουμε με τα συστήματα εγγύησης τραπεζών ε, και με τα ταμεία της εξυγίανσης, ε, προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Αλλά να επαναλάβω, Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε με έναν τρόπο ώστε να πετύχουμε αποτελέσματα και να τα θέσουμε σε εφαρμογή όλα αυτά, γιατί διαφορετικά δεν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε την Ένωση και να τη διατηρήσουμε ενωμένη. Ευχαριστώ. Ο χρόνος πραγματικά πιέζει. Θα ζητήσω από τους να προσπαθήσουν να περιοριστούν σε τρία λεπτάκια. και ίσω οι υπόλοιποι να μην μιλήσουν καν. Θα δούμε. Ελίζα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω το τρίλεπτο. Ουσιαστικά θα παριθμίσω κάποια σημεία. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή μας για το πνεύμα συνεργασίας που ήδη έχει δείξει, γιατί είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και ελπίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση θα είμαστε εξίσου αποδοτικοί και επικοδομητικοί. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2010 ενέκρινε μία συνολική γνωμοδότηση για το πώς θα αντιμετωπίσω μία κρίση συστημικής σε τράπεζες. Νομίζω ότι ήταν σημαντική εκείνη η έκθεση και μάλιστα συγκέντρωσε πλειοψηφία εντασσόταν στο κανόνα 42, στο άρθρο 42 και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια συνέχεια. Τελικά υπήρξαν καθυστερήσεις μεγάλες και άρχισε να φαίνεται κάποια δράση μόνο προς το τέλος της τεράστιας αυτής κρίσης που αντιμετωπίσαμε και μόνο στην τελική φάση ή υπευλήθη μια νομοθετική πρόταση. Βέβαια, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ε, καλωσορίζουμε την πρόταση έστω και αργά και φυσικά θα συνεργαστούμε στην όλη διαδικασία. Θα ήθελα να υπενθυμίσουμε τώρα τους στόχους ε, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για πώς θα διαχειριστούμε μια τράπεζα που αντιμετωπίζει προβλήματα ή μπαίνει σε πτωχευτική διαδικασία. Ε, βασικός στόχος είναι να μειωθεί το συστημικό κόστος ε, μίας ε, μη συντεταγμένης, μη οργανωμένης πτώχευσης. Δεύτερον, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε, να δώσουμε εγγύησει για τις καταθέσεις και για τις τρέχουσες δραστηριότητες. Επίσης, σημαντικό είναι να μην πληρώσουν τα σπασμένα οι φορολογούμενοι να μην πληρώσουν το κόστος μιας ε, τραπεζικής χρεοκοπίας. Επίσης, είναι σημαντικό να διαρρήξουμε επιτέλους το φαύλο κύκλο μεταξύ δημόσιου χρέους και τραπεζικού χρέους. Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι το κυρίως έργο μας. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε σε μια στιγμή που δημοσιεύθηκαν παράλληλα και άλλα κείμενα και άλλες προτάσεις που υιοθετούν μια πιο μέσο και μακροπρόθεσμη προοπτική και που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Μία πρώτη λοιπόν απόφαση που καλούμαστε να λάβουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ είναι να δούμε κατά πόσο στο νομοθετικό αυτό κείμενο θα περιλάβουμε και άλλες διάμεσες αποφάσεις και προτάσεις. Γιατί μερικά από τα στοιχεία της οδηγίας που αναλύουμε δεν συνάδουν πλήρω με μια πιο μέσο και μάκρο πρόθεσμη προοπτική. Μια και δεν έχω χρόνο λοιπόν, θα ήθελα να πω απλώ ότι αναφέρομαι σε κάποια στοιχεία που αφορούν την θέση της 26ης Ιουνίου του 2012 με πρωτοβουλία των τεσσάρων προέδρων για την έκθεση με τίτλο προς μια γνήση Οικονομική και Νομισματική Ένωση και κάποιες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ε, ένα δικό χάρτη προς μια τραπεζική ένωση. Στην, ε, στον δικό αυτό χάρτη περιλαμβάνονται κάποια πολύ κεντρικά σημεία της ε, πρότασης του Ιουνίου των τεσσάρων προέδρων επιτροπών. Οπότε καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη και να εξετάσουμε πρώτα με ποιο τρόπο και ποια οντότητα, ποιος φορέας ή ποια αρχή θα ασχοληθεί με την εκαθάριση μιας τράπεζας. Ιδιαίτερα όταν μια τράπεζα έχει δραστηριότητες σε πολλές ε, χώρες μέλη και έχει και συστημικό χαρακτήρα. Γιατί αυτό το κενό διαπιστώνω εγώ στο κείμενο. Υπάρχει έλλειψη γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό το θέμα. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να έχουμε ένα δίκτυο εγγύησης των καταθέσεων. Με διακόπτετε. Καλώς, εντάξει. Τέλος. I'm sorry. Uh, no... Συγχωρείτε. Δεν ήμουν ευγενική στην αρχή, δεν θα είμαι ευγενική στο τέλος. Επόμενος. Με συγχωρείτε Σάρων, αλλά δεν είναι λογικό. Όλοι είχαν όλο όσο χρόνο θέλανε. Ε, με συγχωρείτε, όχι έτσι κάνουν όλοι. Βολφ Κλίντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι γνωρίζουν πω η πρόταση τη ε, Κομισιόν καθυστέρησε πάρα πολύ. Εμεί θέλαμε να έρθει πολύ νωρίτερα, αλλά ίσω αυτό να είναι καλό γιατί εντωμεταξύ υπάρχουν και νέε σκέψει για την εποπτεία των ε, τραπεζών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάσωση και ένα Ταμείο ε, εγγύηση των Καταθέσεων. Γνωρίζουμε επίσης πως οι τράπεζε είναι το κυκλοφορικό σύστημα της οικονομίας, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργούν ε, σωστά και να μην υφίσταται βλάβε στο υπόλοιπο σώμα της οικονομίας. Νομίζω πως η πρόταση εδώ πέρα έχει αρκετές καλές προσεγγίσεις. Θεωρώ πως η δομή εδώ πέρα, δηλαδή να ξεκινήσουμε τα προληπτικά μέτρα τα οποία θα αφορούν ε, όλες τις τράπεζες οι οποίες θα πρέπει να προετοιμάσουν τα σχέδια λύσης τους και πιθανώς ε, κάποιον ειδικό διαχειριστή για κάποια φάση λύσης ή αναδιάρθρωσης ε, νομίζω πως είναι πάρα πολύ ε, σωστό και παρατηρούμε επίσης πως η Κομισιόν έχει αφιερώσει πάρα πολύ κόπο στο να συμπεριλάβει διάφορες πτυχές που έχουν προκύψει από την πράξη. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλες πτυχές γιατί υπάρχουν και άλλες πτυχές ε, όσον αφορά την πανευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εποπτείας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία και το είπε ο Γκιούνερ για να έχουμε μία ενιαία προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των όσων γίνεται στην Ευρωζώνη και εκτός Ευρωζώνης. Μετά την τελευταία παγκόσμια κρίση είχαμε διαφορετικές ε, προσεγγίσεις ε, και και είναι ευκαιρία να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα, πόσο ορίζουμε το ίδρυμα το οποίο είναι πιθανό να χρεοκοπήσει, να ξεκαθαρίσει η ιεραρχία των διαφόρων περιπτώσεων ε, και το τι γίνεται στα διαφορά μέτρα ή μέσα της ε, λύσης για να μην υπάρξει κάποια στρέβλωση του ανταγωνισμού τα δε μέσα συμμετοχής στην, ε, στις ζημίες ε, των μετόχων θα πρέπει βεβαίως να αφορούν τουλάχιστον να αφορούν, είναι σωστά τώρα το 10% των ε, στοιχείων ενεργητικού είναι το ελάχιστο ή το μέγιστο επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως ο τομέας συνολικά ο χρηματοπιστωτικός πρέπει να προχωρήσει σε μία ε, συγκέντρωση, σε συγχωνεύσεις. Δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στις τράπεζες, ίσως πρέπει να δούμε και ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά ταμεία κτλ. Όλα αυτά είναι χρηματοπιστωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Ε, Φιλίπ. Ευχαριστώ, Φιλίπ. Ευχαριστώ. να επικεντρωθώ στα σημεία που κατά τη γνώμη μου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Καταρχήν, το μέγεθος των ταμείων που θα υπάρχουν στην εξυγίαση. Ε, μιλάμε για 70-75 δισεκατομμύρια μετά από 10 χρόνια, αν κρίνουμε από το ποσό και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που για ένα ταμείο εξυγένσης είναι μάλλον ανεπαρκές, ε, άντε να καλύψει μια-δύο τράπεζες. Υπάρχει περιορισμός λοιπόν σε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, το θέμα του επιμερισμού του κινδύνου. Πόσο ομοσπονδιακή θέλουμε να είναι αυτή η εξυγίαση. Βέβαια γίνεται συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση και νομίζω ότι το θέμα του επιμερισμού αυτού του Resolution Fund, του Ταμείου Εξυγίασης, ξέρουμε ότι είναι τελικά η ίστατη λύση. Ε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει μια, ένας επιμερισμός των ε, διαφόρων ταμείων εξηγένσης μεταξύ των κρατών μελών. Πάντως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις της συζήτησης για την Τραπεζική Ένωση. Ε, μας δεν μας ικανοποιεί και πολύ αυτή η ιδέα. Καλά εγκρίνεται τώρα αυτά που έχουμε επιτάπητος και κάποια στιγμή θα, θα δούμε τι θα γίνει με την Τραπεζική Ένωση. Αν θέλουμε να είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε μια Τραπεζική Ένωση, δεν θα πρέπει να πολλαπλασιάζουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, να χρησιμοποιήσουμε αυτές που έχουμε τώρα για εγγυής καταθήσεων και για την εξυγένση των τραπεζών και να χρησιμοποιήσουμε την νομοθετική διαδικασία για να τι εμπλουτίσουμε με τα σημεία που λείπουν, ώστε να γίνουν μετά και να κάνουμε συμβατή στη συνέχεια την Τραπεζική Ένωση. Αυτή είναι η δική μας θέση και συμμερίζομαι τις ανησυχίες του Βολφ, Κλίντς και άλλων και γνωρίζω ότι ε, το λαμβάνει υπόψη και ο εισηγητής. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε ε, ενιαία την Ένωση, να αποφύγουμε τη διάσπαση και να ε, μην εγκρίνουμε προτάσεις που θα ενισχύουν τον κατακαιρματισμό και τη διάσπαση σε ό,τι αφορά την αρχή της εξυγίασης. Δεν θέλουμε ε, ε, κατακαιρματισμό. Ίσως ε, εμείς είμαστε κατά του φεντεραλισμού. Δεν θέλουμε μια ευρωπαϊκή αρχή να έχει δεσμευτικές εξουσίες. Τώρα, αυτό που λείπει από τις προτάσεις είναι ότι θέλουμε ε, μια κλίμακα παρεμβάσεων. Το κείμενο αυτό δεν προβλέπει απλώς πώς θα παρεύουμε όταν αρχίσουν τα πράγματα και πηγαίνουν στραβά. Να έχουμε ε, και ε, ένα προγενέστερο στάδιο να δούμε πώς μια τέτοια αρχή εξηγήσεις μπορεί να παρέμβει σε ένα ίδρυμα που, βαίνει, που πάει να πάρει το στραβό δρόμο, σε πιο προκαταρκτικό στάδιο. Αυτό, αυτά λοιπόν είναι τα βασικά μου σχόλια. Επαναλαμβάνω, ε, να συνεχίσουμε τις εργασίες ε, με βάση του τι ήδη συζητάτε για την Τραπεζική Ένωση. Βέβαια θα είναι σφοδρές οι συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ομόνια μεταξύ μας από ό,τι στο ΕΚΟΦΗΝ. Και αν κρατήσουμε αυτή την ε, ομόνια και αν προωθήσουμε και τις εργασίες για την τέταρτη οδηγία για την κεφαλαϊκή απέτηση, πιστεύω ότι θα κάνουμε τη διαφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εισηγητής μας εδώ πέρα νομίζω εργάζεται σκληρότερα από όλους και εμείς εργαζόμαστε σκληρά μέχρι την προθεσμία. Προφανώς δεν θέλουμε να χρεοκοπούν ε, οι τράπεζες, θέλουμε τράπεζες που λειτουργούν και μπορούν να δανείσουν στην οικονομία και όταν χρεοκοπεί μια τράπεζα δεν θέλουμε μια τράπεζα κατά τη διάρκεια της κρίσης να ε, βρίσκεται σε κρίση και ίδια. Και να αναγκάζονται άλλοι να μαζεύουν τα σπασμένα. Έτσι καταστρέφεται πάρα πολύ αξία για ολόκληρη την οικονομία. Οπότε πολλά μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε εδώ πέρα. Κάτι το ευρύτερο. Ε, πρέπει η νομοθεσία να είναι σωστή και προ-κρίσης. Εμείς ψηφίσαμε την Οδηγία Κεφαλαϊκών Απτήσεων τον Μάιο και προχτές ε, λάβαμε την πρόταση της Κομισιόν για το συμβασμό για τη ρευστότητα. Αν θέλει όλα αυτά η Κομισιόν να τα κάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, πρέπει να κινητοποιηθούμε λίγο. Μπορεί να έρθει και η Κομισιόν σε κάποιον τριμερή διάλογο εκτός από τους βουλευτές, γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Μάθαμε πως χρειαζόμαστε σχέδια ανάκαμψης και λύσεις, ε, ενδιάμεσα σχέδια, βεβαίως ε, διαγραφή ε, κάποιων απαιτήσεων και βεβαίως κάτι τέτοιο να μην γίνεται μονίμως. Ε, μάθαμε πώς γίνεται αυτό με τα λεφτά των φορολογουμένων και ήταν κάτι το ακριβό και αποτυχημένο. Υπάρχουν και δικαιώματα μετόχων επίσης μέχρι την στιγμή που θα εξαφανιστεί όντως ε, και νομικά η τράπεζα και η ενδο... και η πράξη που γίνονται εντό του ομίλου είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί στην Ευρώπη πηγαίνουν τα λεφτά από τη μία θηγατρική στην άλλη και αυτό πάλι αφορά την οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων και δεν είμαι πάρα πολύ άνετη με τα της μειοψηφίας εκεί πέρα. Αλλά δεν νομίζω πως ε, ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων λειτουργεί για όλα τα κράτη-μέλη, αυτό είναι λάθος. Άλλες χώρες, κάποιες χώρες εξετάζουν την προτίμηση των καταθέσεων για να προστατεύσουν τους φορολογούμενους. Ε, είναι επίσης περίεργο το ότι η πρόταση εδώ πέρα μπλοκάρει την προτίμηση των καταθέσεων καθώς η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε πει στις πορτογαλικές τράπεζες πως έπρεπε να εισαχθεί ή κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν άλλος ένας τρόπος ε, αυτός ε, για το ζήτημα αυτό το σύστημα αυτό εγγύησης καταθέσεων σε άλλες χώρες λειτουργεί ε, μια χαρά. Υπάρχουν βεβαίω και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, και αυτό είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Μια ανησυχεί επίσης η σταδιακή ε, αύξηση αρμοδιοτήτων από παρατηρητής ε, να μεταβληθεί σε ρυθμιστή ποιος και αυτό με απασχολεί στη χώρα μου. Έχουμε και υπερδιατλαντικές μάλλον τράπεζες Παραδείγματο χάρη ε, ήρθε και η Γαλλική Ένωση Τραπεζών που μου είπε πως ε, την απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της εμπιστευτικότητας όταν μιλάμε για τη λύση τραπεζών. Σας ευχαριστώ. Ε, ο χρόνος πιέζει. Από την ΚΟΕ υπάρχει κανείς. Όχι, όχι, ωραία. Πίτερ Ζέιμαν. Α, εδώ είστε. Α, μάλιστα, εντάξει. Ευχαριστώ. Εγώ καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον συγκεκριτή. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ εδώ για να ακούσω την ε, παρουσίασή του. Έπρεπε να πάω σε άλλη επιτροπή για να ψηφίσω την έκθεσή μου. Έτσι λοιπόν, ε, θα αναφέρω μόνο κάποιες από τις ανησυχίες μας και τα πιο γενικά σχόλια για την πρόταση αυτή που έχουμε επιτάπητος. Το πρώτο θέμα, και ζητώ συγγνώμη αν το αναφέραν άλλοι συνάδελφοι, είναι το ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η πρόταση αυτή που συζητούμε δεν εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εξυγένσης των τραπεζών, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά αναχρηματοδότησης, χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν αυτό ε, όπως ξέρετε, εμά θα μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εξυγίανσης ε, και όχι το δεύτερο για προφανεί λόγους. Επίσης, ποιο είναι ο κύριο στόχο του συστήματο αυτό, Ξέρουμε ότι είναι να αποφύγουμε, να είναι οι καταθέτες και οι φορολογούμενοι αυτοί που θα πληρώσουν την ε, κρίση και επίσης ε, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί λοιπόν στο ποιες αναλογίες θα βάλουμε στην ε, εξασφάλιση των καταθέσεων, γιατί θα πρέπει να προστατεύουμε τους καταθέτες και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα είναι σημαντικό να συγκρίνουμε τις διάφορες μελέτες που υπάρχουν ε, για την ικανότητα των ποσών που προβέπονται στην οδηγία σε ό,τι αφορά την ε, ικανότητα απορρόφησης των συνεπειών των σοβαρών κρίσεων. Και κάτι ακόμα έχει να κάνει με την ε, ιεραρχία που παρουσιάζεται στην ε, πρόταση που παρουσιάστηκε το σύστημα της εξυγίασης των πεζών θα χρησιμοποιήσει τους δικούς του πόρους αφού θα έχουν εξαντληθεί ε, το σύνολο της αξίας των μετοχών γιατί εγώ νομίζω ότι θα είναι μια λογική επιλογή αυτή. Και κάτι τελευταίο και μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε ή όχι. Δηλαδή θέλουμε να ξέρουμε αν αρκεί το 1% των καταθέσεων για αυτά που συζητάμε εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, έχει τελειώσει το ωράριο των διερμηνέων και έχουν περάσει και 10 λεπτά ακόμα. Οπότε, εάν συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Ε, ή αυτό, ή δεν θα συνεχίσουμε καθόλου. Με συγχωρείτε. Πίτερ, θέλετε να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Ωραία. Και να με συγχωρείτε. So, try to go in English. Um, the, the proposal we have now uh, brings a link between the deposit guarantee scheme draft of the Commission and